Kollegen. I see that our two Tory fronts want to run again, so there's need. Δύο Tories θέλουν να προβάλλουν πάλι ψηφιότητα και χρειάζονται τις φωτογραφίες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir kommen jetzt zu dem Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε. Πάμε τώρα στην έκθεση για το κοσυφοπαίδιο όπου θα δώσουμε το λόγο στη συνάδελφο Λούνατσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε να καλωσορίσω όλους τους συναδέλφους και τους φιλοξενουμένους που ήρθαν να συζητήσουμε όλοι μαζί. Έφυγαν από την αίθουσα οι Λόρδοι. Μπορείτε να συνεχίσετε γερμανικά. Θα συνεχίσω όμως εγώ παρόλα αυτά αγγλικά, για να μ' ακούνε χωρίς διερμηνία αν ε, έμεινε κανείς. Καλώς ήρθατε όλοι. Ξαναγυρίζουμε στην έκθεσή μου για το κοσυφοπαίδιο που θα συζητηθεί τώρα και θα ψηφιστεί στις 7 Φεβρουαρίου. Ήδη έγινε πριν από κανένα δύο εβδομάδες ε, μια πρώτη συζήτηση, τώρα έχουμε και τις τροπολογίες και είχαμε καλή συζήτηση για τις συμβιβαστικέ με τους Σκιώδης. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους Σκιώδης για την καλή συνεργασία. Ελπίζω να συνεχίσουμε ε, στο ίδιο κλίμα αν χρειαστεί κάποια συμφωνία για το κατάλογο του ψηφοφορία μέχρι τις 7 Μαρτι... Ε, Μαρτίου, είπε, αν χρειαστεί, Φεβρουαρίου θα εννοεί. Ε, λοιπόν, τώρα, τι χαιρετίζουμε στην έκθεση. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που επετεύχθη στην πορεία του Κωσόβου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τις περσινές εξελίξεις, με την προοπτική να αρχίσει φέτος μια συζήτηση για να υπάρχει και συμφωνία σταθεροποίησης και συνεργασίας έχει πληρώσει πολλές προϋποθέσεις στο κοσυφοπαίδιο. Επίσης ε, για τον οδικό χάρτη για τις θεωρήσεις πέρσι δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα επίσης οι αρχές του κοσυφοπαιδίου. Ε, βέβαια πολλά πράγματα πρέπει να δει το Κόσοβο και το θέμα της διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος, καταπολέμησή τους, ανεργία, ε, κράτος δικαίου, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και οικονομικά θέματα. Ε, ε, όπως η ε, ενεργειακά θέματα. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, αλλά πρόοδο βλέπουμε. Και νομίζω ότι εκεί, προς εκεί πρέπει να κινηθούμε, αν και πολλά πράγματα δεν είναι τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση που παίζει ρόλο σε όλα αυτά. Πρόσφατα είχαμε έκθεση ρεμφυγού Συνεδρίου για τη Γιούλεξ, τη μεγαλύτερη μη στρατιωτική αποστολή που έχουμε εκεί και το Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζει την λύπη του διότι πέντε κράτη-μέλη δεν αναγνωρίζουν. Υπάρχει πρόβλημα να συμμετάσχει στην Europol και στην Interpol το κοσυφοπαίδιο, όπου είναι πολύ σημαντικό θέμα η μάχη κατά της διαφθοράς και του εργομένου εγκλήματος. Πολλά θέματα λοιπόν καλύπτουμε και κάναμε συμβαστικές τροπολογίες σε αρκετά θέματα. Ελπίζω να υποστηριχθούν από ευρεία πλειοψηφία σε αυτό το κοινοβούλιο. Να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες που δεν υποστηρίζω, κάποιες που τις υποστηρίζω. Ας δούμε πρώτα αυτές που περιλαμβάνω στις συμβιβαστικές και που θα ε, έχουν θετικό πρόσημο στο δικό μου κατάλογο ψηφοφοριών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες και πολλές ήταν πολύ καλές τροπολογίες σε πολλούς τομείς και τις συμπεριέλαβα ακόμα και τροπολογίε ανθρώπων που ξέρω ότι δεν συμμερίζονται τι δικέ μου ευρείε αντιλήψεις σε σχέση με την κρατική μορφή του Κωσόβου. Οπότε και ε, δέχτηκα αρκετέ τροπολογίες από ανθρώπους που έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας λοιπόν σε αυτό το τομέα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναφερθώ... Α, η φίλη κυρία Κοπά δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι πολλές οι τροπολογίες της και οι τροπολογίες των συναδέλφων της που προσπαθούν... Α, και άλλων συναδέλφων επίσης που λένε ότι δεν είναι κράτος, ε, στην μικ ε, στους αστερίσκους. Όπως ξέρετε δεν δέχομαι αυτές τις τροπολογίες και δεν θα τις ψηφίσω. Και επίσης θέλω να σας θυμίσω ότι ήδη στα δύο προηγούμενα ψηφίσματα εκθέσεις που είχαμε για το κοσυφοπαίδιο ε, ενθαρρύναμε τα πέντε εναπομείναντα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν την κρατική μορφή και την ανεξαρτησία του Κωσόβου. Εμένω αυτό και ελπίζω η πλειοψηφία να συμφωνήσει στο Κοινοβούλιο με μένα. Επίσης, α, θέλω όμως να ευχαριστήσω την κυρία Κοπά και όλους τους άλλους από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που αναφέρθηκαν για παράδειγμα στον αριθμό των χωρών που αναγνώρισαν ήδη το κοσυφοπαίδιο. Δεν το είχα κάνει πριν, αυτό θα το υπερψηφίσω βέβαια και άλλα, άλλα θέματα θα ψηφίσω. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες από συναδέλφους που δεν αναφέρονται σαφώς στην τελευταία εξέλιξη. Η Γιούλεξ έχει τώρα νέα εντολή με σαφώς προσδιορισμένους στόχους και ορόσημα συγκριτική αξιολόγηση. Δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν, τώρα υπάρχει. Υπάρχουν δηλαδή ε, τροπολογίες που θα τις στηρίξω γιατί αναφέρονται σε παραδοθούσες καταστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι κυρία Μπόσκου εδώ, θα τη το πω και προσωπικά. Αναφέρεται στους έργους του Κωσόβου που πρέπει να μπορούν να μιλάνε τη γλώσσα τους παντού στο Κωσυφοπέδιο. Και αυτό πράγματι τώρα υπάρχει στο Σύνταγμα του Κωσυφοπεδίου. Κάθε πολίτης του Κωσυφοπεδίου ε, μπορεί να αξιώνει, να μιλάει και να χρησιμοποιεί την ε, μητρική του γλώσσα σε όλη τη χώρα, σε όλη την επικράτεια. Και ακριβώς γι' αυτό, επειδή έχει αλλάξει τώρα η κατάσταση, δεν ψηφίζει την τροπολογία της. Τώρα, άλλα θέματα ε, σαφώς και συμφωνώ με πολλούς από τους συναδέλφους για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών γίνεται κάποια αναφορά, τη σημασία της ένταξής τους στην ε, κατάρτιση και ανάπτυξη πολιτικών κρατικών. Αυτό βεβαίως και το έλαβα υπόψη. Επίσης πολλές τροπολογίες αναφέρονται σε θέματα κοινωνικά, την ανεργία, τη μεγάλη ανεργία, ε, κυρίως των νέων. Επίσης έχουμε καλή συμβιβαστική τροπολογία για θέματα ε, διάστασης του φύλου, το κοινωνικό φύλο. Ε, υπάρχουν κάποιες καλές εξελίξεις στο Κωσυφοπέδιο. Υπάρχει ένας κανόνας ότι κάθε κόμμα θα πρέπει να έχει το 1 τρίτο των βουλευτών που να είναι γυναίκες και λίγες χώρες το έχουν αυτό και ακόμα λιγότερες το ακολουθούν. Λοιπόν, πολλά καλά, περισσότερα πρέπει να γίνουν ακόμα. Βεβαίως γίνεται αναφορά και στο θέμα του Βορρά και τις τελευταίες μέρες είχαμε πρόοδο με μια συνάντηση μεταξύ των δύο πρωθυπουργών Τάντιτς, Θάτσι την περασμένη εβδομάδα και όλες οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί αλλά υπάρχει πρόοδος και υπάρχει αυτή η έκκληση να σταματήσουν οι αδιαφανείς παράλληλες δομές στο Βορρά, αστυνομία και ε, δικαστική εξουσία και υποστηρίζουμε την ε, κυβέρνηση της Σερβίας ε, και του Κωσόβου για την εκπαίδευση και την υγεία. Αυτά πρέπει να γίνουν σε συνεργασία αγαστή με την κυβέρνηση του, της Πρεστίνα. Η, η πρόοδος στο διάλογο προς τα εκεί κινείται. Εμείς περιμένουμε να δούμε τι έκβαση θα έχουν όλα αυτά. Και σταματώ τονίζοντας κάτι θετικό, το θέμα του διαλόγου τη ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων μεταξύ Σερβίας και Κωσόβου. Εδώ σημειώθηκε καλή πρόοδο. Έχουμε τέσσερι σταθμού συνόρων που λειτουργούν. Την περασμένη εβδομάδα συμφώνησαν για το πώ οι τελωνιακοί δασμοί θα ε, εισπράττονται και θα διανέμονται. Υπάρχει δηλαδή εξομάλυνση στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Παρ' όλα αυτά ξέρω ότι τα πράγματα πρέπει να προχωρήσουν περισσότερο και πολλά περισσότερα πρέπει να κάνει και η ίδια η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου που και είμαστε πολύ επικριτικοί σε σχέση με τις ελλείψεις της χώρας, όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε και τα θετικά που επέτυχαν. Ε, εδώ με αυτή τη θετική νότα κλείνω. Και βεβαίως θα ήθελα και οι συνάδελφοι να τονίσουν και να εστιάσουν περισσότερο στα θετικά στην διαδικασία της διεύρυνσης πρέπει να συμπεριληφθεί και το κοσυφοπαίδιο και γι' αυτό εμείς επικεντρώνουμε στα θετικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόσελτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για την πολύ καλή συνεργασία. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια συνάντηση των σκιωδών με την εισηγήτρια και συμφωνήσαμε απόλυτα επί όλων των συμβιβαστικών τροπολογιών. Βέβαια, επειδή είναι πολλές οι τροπολογίες, ακόμα υπάρχουν σε μερικές διαφορετικές απόψεις. Εγώ συμφωνώ με τη γραμμή πλεύσης της εισηγήτριας για τη σταθεροποίηση της χώρας σε τρεις εβδομάδες έχουμε το πέμπτη επέτειο της ανεξαρτησίας του Κωσόβου και όποιος πάει συχνά στη χώρα αυτή βλέπει τις τεράστιες πρόοδους. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά βάρη ακόμα γιατί υπάρχει ένα ερωτηματικό σε όλα τα θέματα. Και αυτό το ερωτηματικό δείχνει ότι ακόμα υφίστανται δυνάμεις που αμφισβητούν τη χώρα αυτή καθ' αυτή. Αυτό είναι πολύ ε, επικίνδυνο. Αλλαγές συνόρων θα ήταν πρόσκληση για εντελώς καινούργιο καταμερισμό της περιοχής των Βαλκανίων. Και όποιος παίζει κοντά στη Μητρόβιτσα εκεί γύρω με αλλαγές, παίζει και με το Πρέσεβο ε, στο νότιο τμήμα ή στη Βοηβοντίνα Παίζει δηλαδή με την ύπαρξη και την εδαφική ε, ακαιρεότητα της Μακεδονίας, ε, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Γι' αυτό παρακαλώ όλους να ακολουθήσουν το δρόμο τον ευρωπαϊκό. Δηλαδή να μην αποδυναμώσουν την κρατική υπόσταση του Κωσόβου αλλά να την ενισχύσουν. Δεν χρειάζονται υποσημειώσεις εδώ. Η εδαφική ακαιρεότητα να ενισχυθεί, να μην ε, υπάρξουν ε, νέες διαιρέσεις. Τώρα τα σύνορα στην Ευρώπη γίνονται πιο ε, διαπερατά και, όχι, και δεν αλλάζουν. Επίσης προστασία μειονοτήτων όσο γίνεται με περισσότερα ενιαία πρότυπα, προστασία μειονοτήτων στη Μητροβίτσα, στο Πρέσεβο, στο Πρέσεβο δεν υπάρχει ακόμα. Ε, ό,τι ισχύει στο Πρέσεβο πρέπει να ισχύει και στη Μητροβίτσα. Ε, αποφυγή άνισων μέτρων και σταθμών, διπλών ε, προτύπων. Ε, αυτά πρέπει να καταργηθούν. Μόνο έτσι θα σταθεροποιηθεί η περιοχή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό τις ε, μειονότητες στις πολιτικές ομάδες που προέρχονται από χώρες που ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση, βεβαίως θα τις σεβαστούμε, αλλά δεν πρέπει οι μειονότητες αυτές να αποπειραθούν να επιβάλλουν την άποψή τους στην πλειοψηφία. 22 από 27 κράτη-μέλη της Ένωσης το αναγνώρισαν, όλες τις ε, G7 με την, ε, τις ΙΠΑ, Καναδά, Ιαπωνία ε, προχώρησαν στην αναγνώριση εκτός από τη Σερβία όλες οι γειτονικέ όμορες χώρες του Κωσυφοπεδίου αναγνώρισαν την κρατική υπόσταση του Κωσόβου και γι' αυτό παρακαλώ να τεθεί τέλος αυτό το παιχνίδι που συζητάμε εκ νέου κάθε χρόνο για το αν πρέπει να είναι ανεξάρτητο το κράτος. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε ρεαλιστής και στη Σερβία, γιατί έχω πολλές επαφές με Σέρβους πολιτικούς και ξέρουν ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει το κοσυφοπεδίο σερβικό. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έντιμοι και ειλικρινείς απέναντι στους ανθρώπους, στο λαό. Όσο πιο ειλικρινείς, τόσο καλύτερες σχέσεις και πιο γρήγορα θα έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Έχουν γίνει πολλά μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας, αλλά αν αυτά τα θέσουμε ένα αμφιβόλο πάλι, και εμείς θα ευθυνόμεθα για την αστάθεια που θα προκύψει. Ο κ. Παντσέρη. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Λούνατσε και ότι έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά κατά την εκπόνηση των τροπολογιών, των συμβαστικών τροπολογιών και πραγματικά έχει γίνει όλα τα τελευταία χρόνια μια πολύ καλή εξαιρετική δουλειά και βλέπω ότι σήμερα καταβάλλεται μια παραπάνω προσπάθεια προκειμένου να δοθούν κάποιες χρήσιμες ενδείξεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σταθεροποίηση της χώρας προκειμένου να καταφέρει δηλαδή το κοσφοπέδιο να ανταποκριθεί το στομότερο δυνατό στι δεσμεύσει που είχε αναλάβει. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μία συμφωνία σύνδεσης και σταθεροποίησης, γιατί αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει τη μελλοντική ένταξη του Κωσυφοπεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος της EULEX στα πλαίσια της περιοχής αυτής, βάσει της εμπειρίας της οποίας έχουμε ήδη από το παρελθόν. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, ξεκινώντας από τα όσα ήδη λέγονται στην έκθεση του λεκτικού συνεδρίου, που ήδη έχει εντοπίσει κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρχές του κοσμοπεδίου δεν συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία σαφής γραμμή οριοθέτησης προκειμένου να καταλήξει το κοσφοπέδιο με ένα ανεξάρτητο δικαστικό σύστημα. Ήδη μια σημαντική εργασία έχει ήδη επιτευχθεί, σημαντική εργασία όμως πρέπει να γίνει και στο μέλλον από πλευρά κοσφοπεδίου. Ο καθένας βέβαια μπορεί να προσεγγίσει το ζήτημα με διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό όμως να απαγκιστρωθούμε λίγο από το παρελθόν, από την όλη συζήτηση που γίνεται για την εξαρτησία της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια αντικειμενική σύγκληση όλων των πολιτικών δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την έκθεση αυτή και θα ήθελα για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την εισηγήτρια Λούνατσακ. Ευχαριστώ. Κούκαν, Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Έχω διάφορες τροπολογίες και θα ήθελα να σχολιάσω και μερικά σημεία. Πρώτον, κάποιες παρατηρήσεις για την μη αναγνώριση. Όσον αφορά την ενθάρρυνση να αναγνωρίσουν όσοι μέχρι τώρα δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο, νομίζω ότι τέτοιου είδους ενθάρρυνση μπορεί να είναι επικοδοποιητική. Πιστεύω ότι σε διάφορες εκθέσεις και έγγραφα ζητάμε από διάφορες χώρες να κάνουν κάτι, εντάξει, και είναι δικιά τους κυρίαρχη απόφαση να το κάνουν ή να μην το κάνουν. Το άλλο έχει να κάνει με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Η διατύπωση εκεί λέει ότι αυτοί που δεν αναγνωρίζουν πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι αποτελεσματική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους χώρους εκείνους ε, κράτους δικαίου. Εγώ δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την αλήθεια. Είναι υπερβολή. Ή κατά τα άλλα, είναι εξαιρετική, εξαιρετικό τάγραφο πολιτικής αυτό. Θέλω επίσης να στηρίξω την έναρξη των διαπραγματεύσεων όσο γίνεται πιο γρήγορα, SCA, e και ότι έτσι θα μπορέσει το κοσυφοπέδιο να μπει στην, παρετέρω στη διαδικασία ολοκλήρωσης. Τώρα για το διάλογο με τη Σερβία πρέπει να επαναλάβω αυτό που είπα και σήμερα το πρωί όταν συζητούσαμε για τη Σερβία. Νομίζω ότι το δημόσιο, οι θεσμοί πρέπει να ενημερώνονται για τον διάλογο που λαμβάνει η χώρα. Αλλιώς κυκλοφορούν διαδόσεις και οι διαδόσεις και οι φήμες μπορεί να οδηγήσουν σε αμφιβολίες και σε ανησυχίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αντιμετωπίσει η Βαρόνια Άστον. Όσον αφορά τώρα την αποστολή της Γιούλεξ, η Επιτροπή στηρίζει αυτό που γίνεται, αλλά υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Ο επόμενος επικεφαλής θα είναι ο αρμόδιος να τα αντιμετωπίσει αυτά. Και επί τη ευκαιρία αυτή θέλω να στηρίξω ιδιαίτερο στην ερευνητική αποστολή της Γιούλεξ για τους ισχυρισμού που έχουμε στην έκθεση Μάρτιν. Ελπίζω ότι θα οδηγήσει σε αποτελέσματα, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων να έχουμε τα συμπεράσματα για το τι έγινε και τι δεν έγινε. Και όσο πιο γρήγορα το έχουμε αυτό, τόσο το καλύτερο. Ο κύριος Αγκουράκης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καταρχήν πραγματικά ένα οξύμορο σχήμα και νομίζω είναι καθαρό και αποδεικτικό του χαρακτήρα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν συζητάμε για την ένταξη μιας χώρας που έχει αποσχιστεί από μια άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα ε, του Κωσόβου είναι απόσχηση και είναι αποτέλεσμα ενός παράνομου πολέμου του ΝΑΤΟ στην ε, Ιουκοσλαβία και που έχει προκαλέσει όλα αυτά τα προβλήματα με τα οποία ακόμα παλεύουμε. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που υπόθηκε ότι η αλλαγή των συνόρων είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα πρέπει να το αποφύγει κανείς αλλά δυστυχώς αυτό έχει συντελεστεί. Ακριβώς αυτό έγινε με τον πόλεμο του ΝΑΤΟ στην περιοχή και γι' αυτό παιδευόμαστε τόσο πολύ. Ε, δεύτερο ζήτημα, θα ήθελα να σημειώσω ότι οι κυβερνήσει που είναι στις διάφορε χώρε, οι οποίε δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο είναι κυβερνήσει από τα αδελφά σα κόμματα, από τα κόμματα τη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Αν έχετε συνεπώ κάτι να πείτε, να πάτε να πείσετε αυτέ τι κυβερνήσει για το θέμα το ότι δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι άλλα είναι τα ζητήματα που παίζονται και δεν είναι αυτό το θέμα. Τώρα για την έκθεση. Καταρχήν, το βρίσκω εντελώ προσβλητικό για όλες τις χώρες των Βαλκανίων που συζητάμε για την ένταξή τους να, να δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στο θέμα της διαφθοράς όπως γίνεται και εδώ στο σημείο 15. Όχι ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά όταν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα, στη Γερμανία, στη Γαλλία τόση μεγάλη διαφθορά ψηλά, είναι ένα θέμα, είναι υποκρισία να κάνουμε μαθήματα σε άλλους. Και δεν θέλω να επεκταθώ, ξέρετε πάρα πολύ καλά σε τι ε, αναφέρομαι. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανέ ότι αν υπάρχει διαφθορά, αυτή ξεκινάει από τα πάνω. Στην Ελλάδα λέμε το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και άρα σε αυτό το κεφάλι δεν γίνεται απολύτω τίποτα παρά μόνο ε, ευχολόγια. Τέλος, γίνεται λόγος για τη δράση της ε, Γιούλεξ. Ε, εδώ ενηχοποιούνται διάφορα ζητήματα της διαφθοράς για το ότι δήθεν αυτές υπάρχουν επειδή δεν έχει αναγνωριστεί το Κόσοβο. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι Ακριβώ λόγω τη άθλια οικονομική κατάσταση, δυστυχώ η πλειοψηφία τη χώρα είναι αναγκασμένη να ζει σε συνθήκε γκρίζα οικονομία και αυτό θα συνεχιστεί όσο καιρό δεν θα υπάρχουν άλλε καταστάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φανίνκ από την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την Κομισιόν. Πρέπει να πω ότι είμαστε ευγνώμονες ε, προς την κυρία Λούνατσεκ. Συνεργαστήκαμε αρκετό καιρό πολύ καλά μαζί. Είμαστε ευγνώμονες και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο γενικότερα για την υποστήριξη των πρωτοβουλειών μας για το κοσυφοπαίδιο που άρχισαν κυρίως το 2009 και βλέπουμε τώρα τους καρπούς αργά να οριμάζουν ε, η διαδικασία απελευθέρωση θεωρήσεων ανανοέωση των αυτόνομων εμπορικών μέτρων. Δύο παραδείγματα μόνο. Όλοι θα σημείωσαν τα πολλά υποσχόμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων πέρσι το Δεκέμβριο και ιδιαίτερα την αναφορά στην διαδικασία σταθεροποίησης και στη συμφωνία σταθεροποίησης και ε, συνεργασίας. Παρακολουθούμε ε, τα βασικά μεγέθη της χώρας από πολύ κοντά και βέβαια την Άνοιξη θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις αν ε, οι προτεραιότητες αυτές αντιμετωπιστούν σωστά από, τον, από το κοσυφοπαίδιο. Η συγγήτρια Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Θέλω πρώτα απ' όλα να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου προς εσάς συνάδελφοι για όλη αυτή την καλή διαδικασία που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα. Τώρα θα μπω σε λεπτομέρειες, σε ένα δύο σημεία. Το ένα ήταν του κύριου Πόσελτ. Σωστά. Και ευχαριστώ που αναφέρεστε στο γεγονό ότι και σε αυτή την έκθεση το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν έχει υπάρξει διάσπαση ε, της χώρας. Και είναι πολύ καλό που λέτε και τι θα σήμαινε αυτό, όχι μόνο για το Κωσυφοπέδιο, αλλά και για τη Σερβία και για ολόκληρη την περιοχή, τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα. Ευχαριστώ λοιπόν που το λέτε. Τώρα προς τον κύριο Κούκαν. Και σας σας ευχαριστώ για το είπατε. Ξέρω ότι έχετε κάποιες τροπολογίες με τις οποίες θέλετε να βγει η μνήα που έχω συμπεριλάβει εγώ για την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου εκεί που αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει αναγνώριση. Άκουσα ότι σας απασχολεί αυτό και τις σύνδετες τροπολογίες σας. Μέρος αυτών το έχω συμπεριλάβει στις συμβαστικές μου. Παρόλα αυτά, την ε, μνήα για την έλλειψη αναγνώρισης θέλω να το αφήσω. Και το λεκτικό συνέδριο το λέει ξεκάθαρα ότι η συνεργασία, αστυνομίε και τα όλα αυτά θα ήταν πολύ πιο εύκολα αν υπήρχε η αναγνώριση. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά λέω επίσης ότι κύριε Κούκαν και το ξέρετε, ότι η συνεργασία που έχουμε μαζί σας και στην αντιπροσωπεία για την Ανατολική Ευρώπη ήταν πάντα πολύ σημαντική. Θέλω να υπενθυμίσω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για το διάλογο από την κυρία Άστον. Το είπανε και άλλοι και συμφωνώ και εγώ. Θα το ζητήσουμε. Ε, ευχαριστώ και για αυτό που είπατε για τη Γιούλεξ και τον επικεφαλής. όντω, πιστεύω και εγώ ότι θα είναι ο κατάλληλο στη σωστή θέση. Για να πω τώρα και κάτι στον κύριο Γκουράκη, γιατί επικρίνεται σαν υποκριτική την ε, μνήμα στην διαφθορά στο κοσυφοπέδιο που γίνεται στην έκθεση αυτή. Να σας υπενθυμίσω όμως ότι αυτό το κάνουμε σε όλες μας τις εκθέσεις για χώρες όπου υπάρχει διαφθορά. Και φυσικά βεβαίως υπάρχει και διαφθορά σε υψηλό επίπεδο και στις δικές μας χώρες μέλη. Και εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου είχαμε πολύ σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς και το ξέρετε, ο κ. Στάση ήταν μέλος εδώ και ξέρετε ότι καταδικάστηκε σε τετρατή φυλάκιση. Ακριβώς επειδή θέλησε να πάρει χρήματα κάτω το τραπέζι. Βεβαίως και υπάρχει διαφθορά και στις χώρες μας. Αλλά μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Εδώ προσπαθούμε και εγώ πιστεύω ότι και στις χώρες μας πρέπει να το κάνουμε, να το λέμε. Και ακριβώ γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε για τη διαφθορά όταν αυτή λαμβάνει χώρα κι αλλού. Οπότε σας παρακαλώ να μην μιλάτε για υποκρισία όταν αναφερόμαστε στη διαφθορά σε άλλες χώρες, επειδή την έχουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πάντως τους συναδέρφους και τους σκιώδες και όλους και προσβλέπω σε μια πολύ καλή ψηφοφορία στις 7 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Προχωράμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης όπου έχουμε τον κύριο Μιγκαρέλη. Να σας καλωσορίσουμε θερμά. Η συνεδρίαση διεξάγεται μαζί με την αντιπροσωπεία για το Μαγκρέμπ που προεδρεύεται από τον συνάδελφο Παντσέρη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μιγκαρέλη είναι διευθύνων σύμβουλος για τη Μέση Ανατολή και την Νότια γειτονική πολιτική γειτονίας. Θα μιλήσουμε για την κοινή ανακοίνωση για την υποστήριξη της στενότερης συνεργασίας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης στο Μαγκρέμπ με την Αλγερία, Λιβύη, Μαυρετανία, Μαρόκο και την Ισία. Αγαπητέ κύριε Μιγκαρέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντοτε ήθελε την ολοκλήρωση του χώρου Μαγκρέμπ. Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία και ελπίζουμε να αναλυθεί η δράση για την υποστήριξη της περιοχής στη δημοκρατική αυτή μετάβαση και σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο έχουν γίνει πολλά και από μας και έχουν γίνει πολλά και μεταξύ των χωρών αυτών Πολλές φορές ε, ε, η έλλειψη πολυμερών επαφών οφείλεται και για την έλλειψη ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Ελπίζω η κοινή ε, ανακοίνωση να οδηγήσει σε κοινή προσέγγιση προς τις χώρες αυτές με τα προβλήματά τους. Κύριε Μιγκαρέλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματική χαρά να εκπροσωπώ για άλλη μια φορά εδώ πέρα την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να παρουσιάσω την κοινή αυτή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της δικής μου της υπηρεσίας. Πρόκειται για μια παρουσία στην οποία υποστηρίζει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και η ΠΑΤΗ εκπρόσωπος. Για ποιο λόγο θελήσαμε να κάνουμε μια ανακοίνωση που σχετίζεται με τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες του Μακρέμπ. Πολύ γρήγορα θα ήθελα να στις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές. Και τέλος, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντά σα με ποιο τρόπο, κατά την άποψή μα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τι χώρε του Μακρέμπ προκειμένου να αναπτύξουν μια περιφερειακή συνεργασία για να αντιμετωπίσουν καλύτερα από κοινού τι κοινέ αυτέ προκλήσει. Για ποιο λόγο, καταρχά, αυτή η ανακοίνωση. Ο πρώτο λόγο είναι ο ακόλουθο. Οι χώρες του Μαγκρέμπ αποτέλεσαν τις χώρες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή σε, όλες αυτές, σε όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία επηρέασαν την νότια όχθη της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε στην Τινησία, ότι μία από τις χώρες που μετασχηματίστηκε περισσότερο από τα γεγονότα αυτά ήταν η Λιβύη και ότι υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες δεν είχαν ε, μεν επαναστάσεις, αλλά παρόλα αυτά επηρεάστηκαν και γνώρισαν μια πιο βαθμιαία αλλαγή της πολιτικής τους κατάστασης, όπως το Μαρόκο για παράδειγμα ή η Αλγερία. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος ανακοίνωσης είναι ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους οι χώρες του Μαγκρέμπ, οι οποίες αντιμετώπιζαν κάποιες δυσκολίες στη μεταξύ τους συνεργασία, έδειξαν ότι υπήρχαν κάποιες δυνατότητες ε, σύγκλησης, προσέγγισης. Ξέρετε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις οι οποίε δεν είναι πάρα πολύ καλές μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών έγινε μια σειρά από υπουργικέ συναντήσεις ανάμεσα στην Αλγερινή και την Μαροκινή πλευρά που μα επιτρέπουν να πούμε ότι οι δύο αυτές χώρες έχουν καταλάβει ότι πληρώνουν ένα πάρα πολύ ψηλό τίμημα μη συνεργαζόμενες μεταξύ τους και από ό,τι φαίνεται τώρα είναι έτοιμες να συνεργαστούν καλύτερα και βαθμία τελικά να οδηγηθούν σε μια περιφερειακή ολοκλήρωση. Η Τουνησία συνειδητοποίησε το μάθημα αυτό πάρα πολύ καλά. Προσπάθησε μάλιστα να διοργανώσει πέρυσι μια σύνοδο των χωρών του Μακρέμπ, η οποία τελικά όμω δεν διοργανώθηκε. Πάντω, από ό,τι φαίνεται, η Τινήση θα καταφέρουν τουλάχιστον να φέρουν μαζί τους πέντε επικεφαλής ε, των κρατών του ε, Μαγκρέμπα, τους επικεφαλής των πέντε κρατών του Μαγκρέμπ, με Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, ασχολείται ιδιαίτερα με την ανακοίνωση αυτή του Μαρτίου του 2012 όσον αφορά την Αραβική Άνοιξη και θα θέλαμε να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Αραβική Άνοιξη και τις χώρες του Μαγκρέμπ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συντοπίσουμε τις ιδιαιτερότητες των χωρών αυτών. Επίσης η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται και στις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες του Μαγκρέμπ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δηλαδή στο πλαίσιο εκείνο των σχέσεων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αφρικανική Ήπειρο στα πλαίσια της κοινή στρατηγικής Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική. Ένα δεύτερο σημείο τώρα που θέλω να θίξω. Ποιε είναι οι βασικέ προκλήσει τι οποίε καλείται να αντιμετωπίσει η περιοχή του Μαγκρέμπ. Προφανώ εσεί γνωρίζετε τι προκλήσει αυτέ, θα μπορούσα να τι αναφέρω πάρα πολύ γρήγορα. Πρώτον, οι χώρε του Μαγκρέμπ ξεκίνησαν μια διαδικασία εκδημοκρατισμού, η οποία έχει σημειώσει πρόοδο τα τελευταία δύο χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία προ αυτό, αλλά αντιμετωπίζει όλη διαδικασία και κάποια εμπόδια. Ξέρετε ότι στι χώρε αυτέ γίνανε καλές εκλογές. Για παράδειγμα, στη Λιβύη ήταν οι πρώτες εκλογές που γινόντουσαν ποτέ στην ιστορία της χώρας. Για κάποιες άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Τινησία, οι εκλογές ε, για πρώτη φορά γινόντουσαν σε αξιοπρεπείς ε, συνθήκες. Επίσης, ε, η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει ένα νέο ρόλο στις χώρες αυτές οι οργανώσει που εκπροσωπούν του νέου και τις γυναίκες έχουν ενδυναμωθεί, γίνεται μια προσπάθεια προκειμένου το δικαστικό σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό και πιο ανεξάρτητο και εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι γίνεται μια απόπειρα για να δημιουργηθεί μία αντιστάθμιση, μία δημοκρατική δύναμη η οποία θα αντισταθμίσει το πολιτικό καθεστώς στις χώρες αυτές. Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν και κάποια εμπόδια σε αυτή την όλη διαδικασία. Οι φίλοι μας από την Ισία μας λένε ότι εξακολουθούν και υπάρχουν γυναίκες οι οποίες βρίσκονται σε δύσκολη θέση, μάλλον η θέση τους γίνεται ακόμα χειρότερη. Υπάρχουν ορισμένοι καλλιτέχνες οι οποίες αισθάνονται ότι δεν είναι ιδιαίτερα ελεύθεροι Υπάρχουν άνθρωποι οποίοι θα ήθελαν να μπορούσαν να πιούνε κάποια μπύρα ή να πιούνε ένα αλκοολούχο ποτό και τελικά αυτό το κάνουν με όλο και μεγαλύτερη δυσκολία. Βλέπετε ότι αρχίζει και υπάρχει μία πίεση από κάποια συγκεκριμένα κινήματα και κυρίως από τους αλαφιστές Επομένως ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία εκδημοκρατισμού η οποία είναι ουσιαστική και η οποία όμως αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή κάποια εμπόδια. Εμείς τώρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να κινηθούν σε σωστή κατεύθυνση. Η δεύτερη πρόκληση που έχουμε είναι η κοινωνικονομική κατάσταση. Πολύ γρήγορα θα αναφερθώ στο ζήτημα αυτό. Ξέρω ότι κάθε χρόνο υπάρχουν όλο και περισσότεροι νέοι οι οποίοι φτάνουν στην αγορά εργασία, αλλά δεν αυξάνονται αναλογικά και οι θέσει εργασία. Επομένω, αυξάνεται αναγκαστικά η ανεργία συνθήκε διαβίωση δεν έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αντίθετα επιδεινώθηκαν, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μία αναδυόμενη αγανάκτηση στα πλαίσια των πολιτών και ιδίω ανάμεσα στου νέου. Η αγανάκτηση αυτή που όλο και αυξάνεται, αν δεν καταφέρουμε να βοηθήσουμε τι χώρε του Μαγκρέμπ να αναστρέψουν τι τάσει και να οδηγηθούν τελικά σε μια δίκαιη οικονομική ανάπτυξη, τότε η αγανάκτηση αυτή ενδεχομένω από πολιτική πλευρά να μεταφραστεί σε μια επιστροφή σε παρελθούσες στάσεις τις οποίες εμείς θα προτιμούσαμε βέβαια να μην ξαναδούμε σε αυτές τις χώρες. Τρίτη παρατήρηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα γεωργικό. Στις περισσότερες χώρες του Μαγκρέμπ δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα στη Γεωργία λόγω της υποβάθμισης του εδάφους, της ε, μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων, λόγω των κλιματικών αλλαγών. Θέλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε το γεωργικό τομέα και να βοηθήσουμε μια αναδιάρθρωση των γεωργικών δομών, γιατί μιλάμε κυρίως για γεωργικές χώρες, πρέπει να αναλάβουμε δράση προκειμένου να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αναδιαρθρώσουν τη γεωργική τους παραγωγή. Και βέβαια ξέρετε ότι καλούμεθα να βοηθήσουμε την ανάδυση ενός δυναμικού ιδιωτικού τομέα. Ξέρετε ότι στις χώρες αυτές είναι πολύ περιορισμένος ο ιδιωτικός τομέας και η ιδιωτική πρωτοβουλία μολονότι είμαστε υπέρ τη ε, κοινωνική οικονομία τη αγορά, αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε θέσει εργασία, χρειαζόμαστε και έναν ισχυρό ιδιωτικό τομέα, ο οποίο θα μπορεί ελεύθερα να αναπτυχθεί. Ω προ αυτό μπορούμε να κάνουμε ακόμα πολλά πράγματα. Επίση, υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού στι χώρε αυτέ που δεν έχει κοινωνικά δικαιώματα και δεν γνωρίζει κοινωνική περίθαλψη και κοινωνική προστασία. Υπάρχουν πολύ μεγάλε αποκλήσει ανάμεσα στην κοινωνία και από τη μία περιφέρεια στην άλλη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση. Ξέρετε, και το ξέρουμε αυτό αυτό και από τι δικέ μα τι χώρε, ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη αν δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Αυτέ είναι οι βασικέ προκλήσει λοιπόν που αντιμετωπίζουν οι χώρε αυτέ. Και να αναφερθώ πολύ γρήγορα επίση και στι απειλέ εκείνε που βαρύνουν την όλη περιοχή. Θα αναφερθώ κυρίω στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Βλέπετε τι γίνεται τι τελευταίε μέρε στην Αλγερία και στο βόρειο Μάλι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να επισέλθω σε περισσότερες λεπτομέρειες ω προς το ζήτημα αυτό. Τώρα, απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είμαι πολύ σύντομο. Πρώτον, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους περιφερειακούς οργανισμούς τους υφιστάμενους. Υπάρχει η Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ, ο κύριος Μπεναγιάντη είναι ο Γενικό Γραμματέα τη Ένωση αυτή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο πολύ δυναμικό, ο οποίο προσπαθεί να δώσει νέα στην ένωση αυτή, αλλά λόγω της σχέσης Αλγερίας και Μαρόκ βλέπουμε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια έχει γίνει αυτή τη στιγμή από την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ δεν έχει ευοδοθεί. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ να μεταφράσει όλες αυτές τις θεωρητικές μελέτες σε πραγματική ουσιαστική δράση. Έπειτα έχουμε το 5 συν 5, ουσιαστικά την Ένωση εκείνη η οποία φέρνει μαζί την Ιταλία, την Ισπανία, την Γαλλία, την Μάλτα και την Πορτογαλία με τις χώρες, τις αντίστοιχες πέντε χώρες του Νότου. Έγινε τον Οκτώβριο μια συνδιάσκεψη 5 συν 5 στην Μάλτα, έχουν διεξαχθεί πολλές υπουργικέ συνεδριάσεις τους τελευταίους 12 μήνες, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας, των μεταφορών Πρόκειται για ένα φόρουμ ουσιαστικά το οποίο μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Μέχρι στιγμή είναι ένα φόρουμ ανταλλαγή απόψεων απλώ, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε το 5 συν 5 να γίνει ένα φόρουμ με πραγματικέ ουσιαστικέ ιδέε που θα εφαρμόζονται στην πράξη. Και έπειτα έχουμε και την Ένωση για τη Μεσόγειο που μολονότι έχουν καταβληθεί πολλέ γαλλικέ προσπάθειες μέχρι στιγμή ε, μπορούμε να πούμε ότι έχει μια μέτρια επιτυχία. Πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια νέα όθηση και δύναμη στην Ένωση για τη Μεσόγειο και να επιτρέψουμε τελικά στη γραμματεία της Βαρκελόνης να αναλάβει τα μεγάλα αυτά σχέδια τα οποία ξεκίνησαν, όπως για παράδειγμα οι μεγάλοι θαλάσσιοι άξονες ή οι μονάδες αφαλάτωσης στη Λόρδα της Γάζας. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά, πολλά μεγάλα σχέδια τα οποία έχουν ξεκινήσει στα πλαίσια της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε όλες τις περιφερειακές ήδη εφιστάμενες πρωτοβουλίες. Πρέπει επίσης όμως να υποστηρίξουμε και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Σας είπα ότι υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στη διαδικασία αυτή. Ένας λόγος παραπάνω για να αναλάβουμε εμείς δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε δίκτυα κοινωνίας των πολιτών. Η κοινωνία των πολιτών να αναπτύσσεται σε κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά θα ενισχύσουν τη δράση τους και την αποτελεσματικότητά τους μόνο αν καταφέρουν τελικά να συνεργαστούν στα πλαίσια περιφερειακών δικτύων. Οφείλουμε λοιπόν και είναι συμφέρον μας να προωθήσουμε την ε, περιφερειακή αυτή δικτύωση των κοινωνικών, της κοινωνίας των πολιτών. Κάτι ακόμα το οποίο θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για σας που είστε ευρωβουλευτές, θα πρέπει να ενταθούν ε, οι σχέσεις ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των χωρών του Μαγκρέμπ. Ξέρετε ότι σε πολλές από τις χώρες αυτές τα κοινοβούλια δεν δραματίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βοηθήσουμε τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών αυτών προκειμένου να στηρίξουν την κοινωνία των πολιτών. Και μπορούμε να βοηθήσουμε τα κοινοβούλια αυτά αν μοιραστούμε μαζί τους τις βέλτιστες πρακτικές που έχουμε εδώ πέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να δυναμώσουμε λοιπόν τη συνεργασία ανάμεσα σε εσά και αυτούς. Επίσης θα πρέπει να ενδυναμώσουμε επίσης και την ικανότητα, τη διοικητική ικανότητα που έχουν οι τοπικέ αρχέ. Σε ορισμένε χώρε, όπω στην Ιταλία, στη Γερμανία, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στον τομέα τη περιφερειακή τοπική αυτοδιοίκηση. Κάτι αντίστοιχο, στα πλαίσια τη αποκέντρωση, θα πρέπει να γίνει και στι χώρε αυτέ, προκειμένου να οδηγηθούν προ μία καλώ λειτουργούσα αποκέντρωση. Γιατί ξέρω ότι πολλέ φορέ αποκεντρώνουμε, αυτό κοστίζει πολύ ακριβά, αλλά τελικά δεν είναι αποτελεσματικό το εγχείρημα. Σε ορισμένε όμω χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση το εγχείρημα είναι πολύ θετικό και θα πρέπει να το μοιραστούμε μαζί με τι χώρε αυτέ. Επίση, να εργαστούμε με τι χώρε αυτέ στον τομέα των μέσων μαζική ενημέρωση και του πολιτισμού. Ξέρετε ότι οι τομεί αυτοί είναι πάρα πολύ σημαντικοί τομεί για την διάδοση, την περαιτέρω διάχυση τη δημοκρατία και των δημοκρατικών αξιών. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε μαζί του και σε αυτόν τον τομέα. Όσον αφορά τώρα τι παγκόσμιε απειλέ, προφανώ θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί για την καταπολέμηση τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο. Ξέρετε ότι υφίσταται μία κάποια συνεργασία, αλλά δείτε τι γίνεται στην πράξη. Πρέπει προφανώς να κάνουμε περισσότερα πράγματα αν πραγματικά επιθυμούν να επιφέρουμε μία σταθερότητα στην περιοχή αυτή και στην περιοχή νότια του Σαχέλ. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους κινδύνους που έχουν να κάνουν με τα βιοχημικά πυρηνικά όπλα στα έχοντας ένα κέντρο συντονισμού στο Μαρόκο. Έχουμε ξεκινήσει με τέτοια προσπάθεια. Θέλουμε όμως να εντείνουμε τη συνεργασία γιατί θεωρούμε ότι η απειλή αυτή είναι πολύ σημαντική και πάρα πολύ κρίσιμη όχι μόνο για τις χώρες του Μαγκρέπ αλλά και για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε τη μεταρρύθμιση του στρατού, των αστυνομικών δυνάμεων, του δικαστικού συστήματος, προκειμένου να είναι πολύ πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση του εργανομένου εγκλήματος. Πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε κάθε δυνατή προσπάθεια που γίνεται προκειμένου να επιτευχθεί μια πάυση των εχθροπαρξιών και μια συμφιλίωση. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή διονίζονται πάρα, πολλές, πάρα πολλές διενέξεις οι οποίες τροφοδετούν στη συνέχεια την και το οργανωμένο έγκλημα. Στα πλαίσια μια αλληλέγγυα οικονομία θα πρέπει να έχουμε επίση και συστήματα εκπαιδευτικά πιο αποτελεσματικά. Μέχρι στιγμής Υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια στι χώρε αυτές με πολλού πτυχιούχους, αλλά πολλές φορές η ποιότητα κατάρτισης δεν είναι πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν εμείς τα δικά μας υφιστάμενα συστήματα και μέσα για να βελτιωθεί η πανεπιστημιακή και επαγγελματική κατάρτιση στις χώρες αυτές. Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν και πάλι τις χώρες αυτές να δημιουργήσουν περιφερειακά δίκτυα, να κάνουν τις απαραίτητες τεχνικές αλλαγές και να χρησιμοποιήσουν όλα τα προγράμματα υποτροφιών που έχουμε όπως το Tempus, το Erasmus Mundus και το καθεξής. Τώρα στον τομέα των ιδιωτικών, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, νομίζω ότι εδώ πέρα οι στόχοι είναι ξεκάθαροι. Θα πρέπει να καταφέρουν οι χώρες αυτές να έχουν μια πιο ποιοτική παραγωγή, θα πρέπει να βελτιωθούν τα μέσα πρόσβασης ε, σε δανειοδότηση και θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων στην εξωτερική αγορά. Όλα αυτά προφανώς θα πρέπει να γίνουν με μια καλύτερη εστίαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ουσιαστικά είναι αυτές που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της οικονομίας και θα δημιουργήσουν τις μελλοντικέ θέσεις εργασίας που χρειάζονται οι χώρες αυτές. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μετέχουν περισσότερο στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την έρευνα, ιδίω το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, πολύ σημαντικό για αυτές τις χώρες, και θα πρέπει να δημιουργήσουμε και δίκτυα μεταξύ επιχειρηματιών, να δημιουργήσουμε επίσης δίκτυα πρόσβασης σε παροχή συμβουλών προς τις επιχειρήσεις των χώρων αυτών. Στον εμπορικό τομέα θα πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη εμπορική ολοκλήρωση των χωρών του Μαγκρέμπ μεταξύ τους και θα πρέπει αυτή η περιφερειακή ολοκλήρωση να ενταχθεί στις ζώνες ελεύθερων συναλλαγών που προσπαθεί να θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Είναι σαφές όμως θα είναι πολύ δύσκολο να βοηθήσουμε ή να πετύχουμε την οικονομική περιφερειακή ολοκλήρωση του Μαγκρέμπ όσο θα είναι κλειστά τα σύνορα μεταξύ Μαρόκου και Τινησίας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε Μαρόκου και Αλγερίας, με συγχωρείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα τα οποία έχουμε εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό. Στον τομέα των μεγάλων δικτύων πιστεύω ότι θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στον τομέα της ενέργειας και της μεταφορές. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο μεταφορών, ιδίως όσον αφορά τις οδικές μεταφορές και όσον αφορά τους αυτοκινοδρόμους ανάμεσα στις χώρες του Μαγκρέμπ και να δημιουργηθεί και ένας εναέριος χώρος ευρώ μεσογειακός. Θα πρέπει επίσης οι χώρες αυτές να αναπτύξουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να γίνουν πιο απαιδευτικές από ενεργειακής πλευράς και θα πρέπει να ενταχθεί η δική τους αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στη δική μας την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλές δραστηριότητες ήδη έχουν ξεκινήσει, αλλά θα πρέπει πάλι να επιταχύνουμε εδώ πέρα και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας. Υπάρχει ένας ακόμα τομέα με τον οποίο θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί τους, γιατί πρόκειται για μια πραγματική απειλή όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το περιβάλλον ουσιαστικά και με τις κλιματικές αλλαγές. Οφείλουμε να συνεργαστούμε με τις χώρες αυτές, γιατί ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού, των θαλασσίων πόρων, Καταλαβαίνετε, στου τομεί αυτού έχουμε πολλά κοινά συμφέροντα και θα πρέπει να ενταθεί η συνεργασία και ο σχετικός διάλογος. Στον τομέα τέλος της προστασίας των πολιτών θα πρέπει να εντείνουμε και στον τομέα αυτό τη συνεργασία μας γιατί υπάρχουν διάφορες φυσικές καταστροφές ανθρωπογενείς οι οποίες λαμβάνουν χώρα στις χώρες αυτές και έχουν επιπτώσει όμως και σε εμά και το αντίστροφο. Οφείλουμε λοιπόν και στον τομέα αυτό να συνεργαστούμε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο κύριε Πρόεδρο, ολοκληρώνω στο σημείο αυτό. Προφανώς όμως κάλυψε ένα πολύ μικρό μόνο τμήμα των προτάσεων που γίνονται στην ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΥΠΑ της εκπροσώπου. Σας ευχαριστώ. Ehm, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Μιγκαρέλη για την παρουσίαση αυτή που έκανε και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μία δράση για να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την περιοχή αυτή στην φάση του εκδημοκρατισμού στα πλαίσια πολυμερών αλλά και διμερών δράσεων και σχέσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουμε πιο κοντά στις χώρες αυτές του Νότου της Μεσογείου. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ανακοίνωση αυτή να υπογραμμίσουμε μια πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να αναφερόμαστε απλώ σε ένα γενικό κατάλογο παρεμβάσεων μπορούμε να κάνουμε για την καλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση του Μαγκρέμπ. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει πραγματικά να ανταποκριθούμε σε μια πολιτική πρόκληση. Γιατί αν δεν το πετύχουμε αυτό το πράγμα, διαφορετικά θα καταλήξουμε τελικά με ένα έγγραφο το οποίο στην πράξη δεν θα πετύχει του αναμενόμενου στόχου. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκεφτούμε το ακόλουθο η περιοχή αυτή διανύει μια τέτοια συγκυρία η οποία απαιτεί πολύ γρήγορες αντιδράσεις από τις υπηρεσίες της ΥΠΑ της εκπροσώπου, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της ασφάλειας ή στο ζήτημα του Μάλι. Καταλαβαίνετε ότι η επικαιρότητα στους τομείς αυτούς επιβάλλει την ανάληψη δράσης. Ήδη στην έκθεση Πιόννα που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κάνει ήδη έναν κατάλογο δράσεων που θα έπρεπε να αναλυφθούν προκειμένου να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε τις χώρες του Μαγκρέμπ. Το κείμενο λοιπόν αυτό, το χαιρετίζουμε προφανώς, είναι πολύ θετικό, αλλά φτάνει ουσιαστικά με δύο χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επομένω, πρέπει να δούμε αν πραγματικά είναι συνεκτική η δράση μα και αν όντω θα καταφέρουμε τελικά να ανταποκριθούμε γρήγορα στι ανάγκε που έχουν οι χώρε αυτέ. Να προσθέσω κάτι ακόμα. Το ζήτημα της περιφερειακής ολοκλήρωσης αποτελούσε ήδη έναν στόχο της διαδικασίας της Βαρκελόνης του 1995 που προέβλεπε τότε τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών το 2010. Δείτε πόσο χρόνο έχουμε χάσει και πόσα προβλήματα στο ενδιάμεσο διάστημα θα μπορούσαμε να είχαμε επιλύσει. θα μπορούσαμε να έχουμε εκμεταλλευτεί επίση και τι ευκαιρίε που μα δίνονται από την Αραβική Άνοιξη. Αν πραγματικά όμω θέλουμε τώρα να ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο, το λέει και η ίδια η έκθεσή σα, η ανακοίνωση αυτή, ότι θα πρέπει οι χώρε του Μαγκρέμπ να αναλάβουν οι ίδιες δράσεις για να στεφτεί με επιτυχία η περιφερειακή ολοκλήρωση, από μόνοι τους δηλαδή να το πετύχουν. Πρέπει προφανώς και η Ευρώπη όμως να συμβάλλει και θα πρέπει να διδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν θα πρέπει όμως να απευθυνόμαστε μόνο στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις κοινωνικές οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, που γνωρίζουν καλύτερα τελικά οι οργανώσεις αυτές ε, ποιε είναι οι απαιτήσει οι οποίες υφίστανται για μια καλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση στη ζώνη αυτή. Και είναι πολύ σημαντικό η πολιτική συνεργασία που βρίσκεται στο κέντρο της δράσης μας και η οποία αναφέρεται στο κείμενο αυτό, να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικού διαλόγου. Και αυτό προσπαθούμε εμείς να προωθήσουμε μέσω των διακοινοβουλευτικών συνεδριάσεων που κάνουμε. Και προσπαθούμε στα πλαίσια της ευρωμεσογειακής σχέσης, με όλες τις πτυχές, οικονομική, περιβαλλοντική, να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό. Όλες όμως αυτές οι δράσεις θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια σε ένα θεσμικό πλαίσιο ξεκάθαρο, όπου θα είναι ξεκάθαρε οι αρμοδιότητες και ευθύνε του καθενό. Δεν θα πρέπει ο καθένα να κάνει ό,τι θεωρεί ότι είναι σκόπιμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να συντονιστούν μεταξύ του. Είναι θετικό δηλαδή το ότι στο κείμενο λέγεται ότι πρέπει να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία και καλύτερε συνταλλαγέ μεταξύ των κοινοβουλίων των χωρών του Μαγκρέμπ και των Εθνικών Κοινοβουλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόλον ότι αυτό λέγεται και είναι θετικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ενισχυμένη συνεργασία να γίνεται στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου και με έναν καλύτερο συντονισμό. Πρέπει επίσης να πούμε ότι Απέναντι στην κατάσταση αυτή την οποία βλέπουμε στο Μάλι και στην περιοχή αυτή θα πρέπει να υπάρχει και μία συνάντηση, μία συνεδρίαση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των χωρών του Μαγκρέμπ προκειμένου η μονομερής αυτή τη στιγμή στρατιωτική δράση που υπάρχει επί τόπου να συνολευθεί και από μία πολιτική δράση Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να πετύχουμε την ευκταία αυτή σταθερότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια τη οικονομική πολιτική που θέλουμε να προωθήσουμε στα πλαίσια τη περιφερειακή ολοκλήρωση. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα θεμελιώδε, να συνεχιστεί ο διάλογο με όλου του συνομιλητέ μα, με τι αντιπροσωπείε που έχουμε για τι χώρε του Μαγκρέμπ, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να γίνει και ένα η ύψιστος πολιτικός διάλογος με την Ένωση του Ραβικού Μαγκρέμπ. Έχουμε προωθήσει και εμεί στο παρελθόν την πρόταση αυτή. Χθε, όπως είπε και ο κύριο Μιγκαρέλη, ο Επίτροπος Φούλε και ο Γενικό Γραμματέας της Ένωσης αυτής συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να συζητήσουν τις προτάσει αυτέ που γίνονται στην κοινή ανακοίνωση και αναφέρθηκα να δεν κάνω λάθος, σε κάποιες πρωτοβουλίες στον τομέα της ενέργειας, στην ε, δημιουργία του ιδιωτικού τομέα, στον τομέα των μεταφορών, στην ε, τομέα της ανάπτυξης ε, της γεωργικής και της υποστήριξης κοινωνίας των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει και η απαραίτητη πολιτική πλέον συνεργασία στο περιβάλλον αυτό το οποίο συνεχώς αλλάζει. Και ελπίζω λοιπόν ότι η δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποτελέσουν στο μέλλον πτυχές μιας κοινή δράσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν στο κείμενο αυτό να μην παραμείνει με ένα θεωρητικό κείμενο, αλλά ένα κείμενο το οποίο θα οδηγήσει σε έμπρακτη δράση επιτόπου. Κολέγκα ε, Η κυρία Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μιγκαρέλη για την παρουσίασή του, όπως πάντα ήταν ιδιαίτερα πλήρης και ορθή. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί δυσκολευόμαστε να θέσουμε σε εφαρμογή όλη αυτή την λεπτομερή παρουσίαση που μας έκανε. Αυτό το όραμα που μας παρουσίασε και που αναμφίβολα ανταποκρίνεται στις ανάγκες για δική μας συμμετοχή και διάλογο με τις διάφορες πλευρές της κοινωνίας των χωρών νοτίως της Μεσογείου. Θέλω επίσης να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Αναφερθήκατε στα εμπόδια για τη δημοκρατία που έχουν να κάνουν ε, σε ένα βαθμό με την άνοδο του κινήματος των σαλαφιστών στις χώρες αυτές. Σε πολλές χώρες είναι η ανεργία, η ανεργία των νέων που παίζει ε, σημαντικό ρόλο και κάνει την ανεργία να αυξάνει. Υπάρχουν χώρες όπου δεν υπάρχουν σύνταξες, στη Λιβύη για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν τέτοια προβλήματα που έχουν να κάνουν ε, με το Κατάρ ε, κλπ. Δηλαδή φεύγει ο κόσμος και πηγαίνει σε τέτοιες χώρες. Τι κάνει λοιπόν η κυρία Άστον για τις χώρες εκείνες οι οποίες ενισχύουν τέτοιου είδους κινήματα τα οποία έχουν τόσο αρνητικές επιπτώσεις. Το στοιχείο τζιχάτ, τρομοκρατία γιατί λοιπόν προκαλείται, από πού. Τα τόσο σοβαρά πρόσφατα γεγονότα που είχαμε στην Αλγερία εξαιτία της κρίσης στο Μαλί. Εσείς πώς τα αναλύετε, πώς αναλύετε δηλαδή αυτά που έγιναν. Και δεν σας ζητάω να αναφερθείτε στην αγριότητα του εγχειρήματο. Εντάξει, υπάρχουν ένα σωρό εξηγήσει γι' αυτό. Υπάρχουν όμω πηγέ. Εγώ είχα επαφέ με μέλη από την αντιπολίτευση τη Αλγερία, οι οποίοι πιστεύουν ότι αυτά τα οποία έγιναν, δεδομένου μάλιστα ότι δεν οργανώθηκαν από τη μια στιγμή στην άλλη, ήταν πράγματα που μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει. Έχουν να κάνουν με εσωτερικές διαμάχες στην Αλγερία ένα παιχνίδι δηλαδή που παίζεται εκεί. Οι αλγερινές αρχές, κατά τη γνώμη σας, τι κάνουν στη χώρα, τι προκαλούν. Η κοινωνία σε τι κατάσταση βρίσκεται τότε. Δεν υπάρχουν κινήματα πολιτών στην Αλγερία είναι κάτι το οποίο επιδεινώνει την κατάσταση και επιτρέπει τέτοιου είδους επικίνδυνες καταστάσεις να δημιουργούνται. Είτε πρόκειται για τρομοκρατία, είτε πρόκειται για διάφορες μαφίες που δρούν. Με τον κίνδυνο CBRN που αναφέρατε κι εσείς. Στην Λιβύη δεν υπάρχει στρατός, η άλλη δύναμη που να μπορέσει να προστατεύσει μία αντίστοιχη μονάδα φυσικού για παράδειγμα και ο κόσμος τρέμει εκεί. Κανένας τελικά δηλαδή δεν ελέγχει την επικράτεια της Λιβύης. Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα είπατε ότι η επίλυση διαφορών έχει τεράστια σημασία. Υπάρχει μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκο διαμάχη, υπάρχει η διαμάχη του Σαχέλ. Εγώ το είδα, πήγα επί τόπου και είδα ότι το αποτέλεσμα είναι να μαζεύεται κόσμος και να προσχωρεί σε διάφορες συμμορίες. Ξέρω την ιστορία, ξέρω ότι είναι διχασμένος ο κόσμος, αλλά όταν μπορούμε να δούμε τον κίνδυνο τη στιγμή που οι τρομοκράτες αυτό ακριβώς θέλουν για να μπορέσουν να πάρουν στις τάξεις του όλο και περισσότερο κόσμο. Είτε πρόκειται λοιπόν για τη Δυτική Σαχαρά, είτε πρόκειται για το Μαλί. Είναι δυνατόν να εξακολουθούμε να κλείνουμε τα μάτια. Αυτά. Και εγώ έχω να ρωτήσω μερικά πράγματα, λέει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Αναφερθήκατε στο ζήτημα της συνεργασίας στα πλαίσια των χωρών του Μαγκρέμπ. Και σίγουρα η πρόκληση αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη γιατί οι χώρες αυτές διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Αίγυπτος, Μαρόκο, Λιβύη, την Ισία διαφέρουν πάρα πολύ και έχουν και διαφορετική ιστορία η κάθε χώρα. Παρ' αυτά αναφερθήκατε σε κάποια μέσα με τα οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η ολοκλήρωση. Αναφερθήκατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διπλωματία, στον πολιτισμό, σε επαφές μεταξύ των κοινοβουλίων. Θα ήθελα λοιπόν να σα ρωτήσω το ακόλουθο. Ποια είναι η άποψή σα για μία συνεργασία στα πλαίσια των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δραματίσει ένα σημαντικότατο ρόλο στην ε, δημιουργία των δικών μας ευρωπαϊκών συστημάτων πρόνοιας. Έχουν βοηθήσει τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Δεν θεωρείται λοιπόν ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα, μη, ένα μέσο όχι μόνο οικονομικής αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης. Μία ακόμα ερώτηση. Ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα, δύσκολη ερώτηση αυτή, ποια είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την καταπολέμηση της τόσο εκτεταμένης διαφθοράς που βλέπουμε στις χώρες του Μαγκρέπ, κυρίως στην άρχουσα τάξη, στην κυβέρνηση και που ουσιαστικά βρίσκεται πάρα πολύ μακριά από τους πολίτες και δημιουργεί τεράστιες ανισότητες και επίσης αλλάζει και στρεβλώνει τους κανόνες της αγοράς και ουσιαστικά καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την επιχειρηματικότητα, ιδίω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και να φέρουμε κυρίως περιοχέ περιοχές εκείνες που δεν υπάρχει μια κάποια κυβερνητική σταθερότητα. Εσείς αναφερθήκατε στις επαφές και το διάλογο ανάμεσα στα κοινοβούλια. Συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση αυτή. Θα μπορούσαμε όντω να εργαστούμε έτσι. Θα πρέπει όμω να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ ανάμεσα στα κοινοβούλια τα κοινοβούλια των χωρών αυτών έχουν μια πολύ νοπή, αν θέλετε, ακόμα πολύ πρόσφατη εμπειρία της δημοκρατίας. Επομένως, οι βουλευτές των χωρών αυτών δεν έχουν τις αρμοδιότητες και την εξουσία που έχουμε εμείς, βουλευτές και ευρωβουλευτές στην Ευρώπη. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προσδώσουμε στους ανθρώπους αυτούς, να τους μεταδώσουμε την δική μας την εμπειρία στα πλαίσια της αποκέντρωσης. Πώς μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να αναλάβουν περισσότερη εξουσία σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Αναφερθήκατε σε αυτό και αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Ιταλίας και άλλων χωρών. Αυτό είναι μια άλλη μορφή δημοκρατίας και διακυβέρνησης. Θα πρέπει όμως τόπου να υπάρχει και μια διαφορετική ποιότητα διακυβέρνησης. Γιατί αν διαβιβαστούν εξουσίες και κονδύλια σε χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο, αλλά εκεί πέρα δεν υπάρχει απαραίτητη ποιότητα διακυβέρνηση, τότε πραγματικά μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια απόλυτη αναποτελεσματικότητα διακυβέρνηση και σε επιζήμιε επιπτώσει για του πολίτε. Ολοκληρώνω τέλο αναφερόμενο στι επιχειρήσει, στου επιχειρηματίε. Ξέρετε ότι κανένας επιχειρηματίας δεν πρόκειται να επενδύσει σε μία περιοχή αν δεν υπάρχει ασφάλεια, κράτος δικαίου και σωστές προϋποθέσεις ε, εμπορικές, οικονομικές. Το να μιλάμε για επιχειρηματικότητα και προώθηση της ιδιωτική πρωτοβουλίας χωρίς να έχουμε επιλύσει πρώτα τις βασικές αυτές προϋποθέσεις καταλαβαίνετε ότι καθιστά όλο το εγχείρημα ιδιαίτερα πολύπλοκο. Ευχαριστώ. Madame vous ε, Ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαγκρέπ είναι ζωτική σημασία. Οι κοινωνίες αυτές βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Οι συζητήσεις που γίνονται στο Μαγκρέπ είναι ίδιες που γίνονται και εδώ στην Ευρώπη. Δηλαδή τι είδου κοινωνία θέλουμε, τι είδου ελευθερίες, ποιο είναι ο ρόλος ε, της κοινωνίας, της θρησκεία κλπ. Γι' αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη Υπάρχουν δύο δυνατότητες μια εναλλακτική για την νεολαία, η οποία ζει άσχημα, είναι απελπισμένη, με τεράστια ανεργία, με φτώχεια. Η εκπαίδευση έχει σημασία, το επίπεδο της παιδείας. Εμείς που είμαστε από τη Μεσόγειο, ακριβώς επειδή είναι γειτονέ μας, επειδή ιστορικά έχουμε δεσμούς κτλ, κάνουμε. Μάλλον θα θέλαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν το κάνουμε όμως. Λοιπόν, ή που θα έπρεπε να το κάνουμε ή που αν δεν το κάνουμε, τότε οι νέοι θα στραφούν αλλού και θα γίνουν ε, θύματα υποχείρη διαφόρων κινημάτων, είτε πρόκειται για την Τσιχάντ, είτε πρόκειται για οτιδήποτε, που στηρίζουν χώρες όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία. Χώρες που παίζουν σημαντικό ρόλο αρνητικό όμως. Στηρίζουν ορισμένα κόμματα και όχι άλλα ότι κυκλοφορούν βίντεο με την άποψή τους για μια κοινωνία κλειστή ε, που πάει πίσω αντί να πηγαίνει μπροστά. Η νεολαία λοιπόν πρέπει να είναι στο κέντρο της δράσης μας. Η νεολαία είναι αυτή η οποία περιμένει από εμά, είναι ανοιχτή, κοιτάζει τα κοινωνικά δίκτυα, κοιτάζει τηλεόραση, την ευρωπαϊκά κανάλια επίσης. Μέχρι τώρα ήμασταν απόντες. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε, να τίνουμε χείρα ε, βοηθείας, αλλά σεβόμενοι μια σχέση ισότιμη μαζί τους. Το πρόβλημα με την Μεσόγειο είναι ότι οι σχέσεις μας βασίζονταν σε πυλώνες που δεν ήταν αρκετά στέρεοι. Και τι ήταν, ήταν η ιδέα ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα θέλουμε νέες αγορές για τις οικονομίες μας και αυτές θα τις βρούμε σε εσά στο Νότο. Δηλαδή είδαμε την Μεσόγειο σαν μια νέα αγορά που θα βοηθούσε τις οικονομίες μας. Με ένα παράδεκτο κάτι τέτοιο. Λέω ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή που πρέπει να κάνουμε επιλογές για το τι κοινωνία θέλουμε. Κάτι που πιστεύω ότι είναι σημαντικό είναι το θέμα της εκπαίδευση και του πολιτισμού. Η Ένωση του Μαγκρέπ. Κοιτάξτε, η ιδιαιτερότητα των κοινωνιών αυτών είναι ότι δεν είναι ακριβώς αραβικές μόνο. Είναι και οι Βερβέροι. Οπότε το να μιλάμε για ένωση του αραβικού Μαγκρέμπ, γιατί αυτό είναι ο επίσημο τίτλο, δεν είναι καλό. Ούτε για του Βεβέρους, ούτε για του Ταμαζάκ μιλάμε, λες, και δεν είναι από εκεί. Πρώτο θέμα λοιπόν, πλουραλισμό. Υπάρχει ένα φιλόσοφο, ο Χατιμπή που πέθανε πριν από λίγα χρόνια και που το βρίσκω καταπληκτικό, έχει γράψει ένα βιβλίο που μιλάει ακριβώς για τον πλουραλισμό στο Μαγκρέμπ. Ο πλουραλισμός είναι πολύ σημαντικός. Αν τον αναγνωρίσουμε, κάνουμε σφάλμα. αν το δεχτούμε, δεχτούμε τον πλουραλισμό στον πολιτισμό, στη γλώσσα. Μπορεί κανείς να είναι μουσουλμάνος. Υπήρξαν πάντα και χριστιανοί και Εβραίοι στη περιοχή. Είναι βασικό λοιπόν να δεχτούμε και να σεβαστούμε τον πλουραλισμό αυτό και να προσέξουμε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους από την περιοχή αυτή, να τις χτίσουμε ακριβώς πάνω σε αυτό τον πλουραλισμό. Τώρα, κατά τα άλλα, ο προλαλής σας αναφέρθηκε στη διαφθορά και στο θέμα του δικαίου. Μα είναι ζωτική σημασία. Πάρα πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν θέλουν να επενδύσουν επειδή νιώθουν ότι δεν υπάρχει νομική ασφάλεια. Αν υπάρξει κάποια διένεξη στην Αλγερία δεν πρόκειται να το λύσετε μέσω των δικαστηρίων. Άρα το θέμα της δικαιοσύνης και μιας στέρεας ε, ε, βάσης δικαιοσύνης είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει στις συνομιλίες μας. Κάτι άλλο το οποίο με ενόχλησε και εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή είχε να κάνει με την κατάργηση των δασμών. Σε όλες τις ε, σχέσεις και συμφωνίες απαιτούμε κατάργηση των δασμών από του εταίρους μα, παρόλο που μερικέ φορέ βρίσκονται σε πάρα πολύ ευάλωτη θέση. Είναι σφάλμα να πετούμε κάτι τέτοιο, γιατί κάνει τι ήδη ευάλωτε οικονομίε του ακόμα πιο ευάλωτε. Επανέρχομαι στην νεολαία, που πρέπει να είναι στο κέντρο των ενδιαφερόντων μα και τι σχέσεις μας μαζί με τις χώρες αυτές. Πρέπει να ακούσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να έχουμε σχέσεις και να ακούμε όχι μόνο ε, τις ηγεσίε αλλά τις κοινωνίες των πολιτών γιατί οι μελλοντικοί ηγέτες θα προέρθουν ακριβώς από εκεί. Τέλος. Για την κοινωνία των πολιτών υπάρχει ένα κοινωνικό φόρουμ ε, από το Μαγκρέπ που βοηθάει και την προετοιμασία του Παγκόσμιου Φόρουμ που θα γίνει στην Ισία το Μάρτιο του 2013 και μπορούμε μέσα από εκεί να γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα τις κοινωνίες των χωρών του Μαγκρέπ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βένσον έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ κύριε Βένσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και για τις εξαιρετικές πληροφορίες που μας δώσατε. Θέλω να αναφερθώ στην νησία που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ίσως δεν κατάλαβα καλά, αλλά ήμουν πολύ προσεκτικός. Μιλήσατε για ισότητα ευκαιριών που έχει αποδυναμωθεί στην Τινησία, είπατε. Ε, από την άλλη έχει μια ιδιαιτερότητα η Τινησία σε σχέση με τις άλλες χώρες. Ε, υπάρχουν ε, πολλοί σπουδαστές και ε, στα μέσα ενημέρωσης επίσης ε, και πολλές γυναίκες. Έτσι λοιπόν, πώς επιδεινώθηκε η κατάσταση των γυναικών στην Τινησία. Ο τουρισμός πάντα έπαιζε στο παρελθόν τεράστιο ρόλο για τη χώρα αυτή. Σήμερα τι ρόλο παίζει ο τουρισμός στην Τινησία. Ευχαριστώ. Vous Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ με όσα είπατε κύριε Πανσέρη για παράδειγμα για την αναγκαιότητα να εφαρμόσουμε συγκεκριμένα όλες αυτές τις ωραίες ιδέες. Όντως δεν πρέπει όλα αυτά να μείνουν σε ένα σιρτάρι. Έχετε δίκιο. Κύριε Γκόμες, βγήκε όμως. Ρώτησε διάφορα πράγματα. Θα απαντήσω πρώτα στα δικά σας, στο μεταξύ μπορεί να επανέλθει κύριε Γκόμες. Δεν θα ήταν χρήσιμο τις εμπειρίες μας για τα συνδικάτα, λέτε, να τις ε, συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε μεταξύ μας. Φυσικά, όταν μιλάμε για την κοινωνία των πολιτών, μιλάμε για τις ε, οργανώσεις, τις ε, διάφορες μη κερδοσκοπικές, αλλά μιλάμε και για τα συνδικάτα. Εννοείται, ασφαλώς. Στην Τινησία, για παράδειγμα, το συνδικάτο το οποίο είναι ισχυρό, η ΙΖΕΣΕ, e, είναι ένα συνδικάτο που παίζει σημαντικό ρόλο και με τα δικά μας τα συνδικάτα και με το, τις δικές μας εμπειρίες από το συνδικαλιστικό κίνημα βοηθάμε τις χώρες αυτές να αναπτύξουν τα συνδικάτα τους. Συμφωνώ μαζί σας και μάλιστα ίσως θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή μήπως μπορεί να θέσει σε επαφή τα συνδικάτα μας με εκείνα των χωρών αυτών. Πολύ καλή ιδέα. Δεν το λέμε ρητά στο κείμενό μας, αλλά ισχύει. Άλλο θέμα. Πώς καταπολεμάται η διαφθορά πρέπει να υπάρξει ο έλεγχος ε, πρώτα απ' όλα της ηγεσίας, γιατί αν η ηγεσία είναι μέσα στη διαφθορά πώ θα καταπολεμήσει τη διαφορά των άλλων. Και χρειάζεται και ανεξάρτητη δικαιοσύνη βέβαια. Σε αυτό πρέπει να του βοηθήσουμε. Ανεξάρτητη δικαιοσύνη και μέσα ενημέρωση είναι δύο θέματα στα οποία του βοηθάμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε αποτελεσματικοί, αλλά ξοδεύουμε εκατομμύρια ευρώ στα διάφορα προγράμματα αρρωγή που έχουμε μαζί του για να του καταρτήσουμε σε θέματα δικαιοσύνη και για να του βοηθήσουμε να αναπτύξουν ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση. Ελπίζω να έχουμε κάποια επίδραση θετική σε αυτό. Οπότε να μπορέσουν να καταπολεμήσουν και τη διαφθορά πιο αποτελεσματικά. Τώρα η κοινωνία των πολιτών βέβαια και στι δικέ μα τι χώρε, παίζει σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση τη διαφθορά. Οπότε αν βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε να έχουν μια ισχυρή κοινωνία των πολιτών θα τι βοηθήσουμε και να αντιμετωπίσουν τη διαφθορά. Αποκέντρωση τώρα και κίνδυνη τη. Έχετε δίκιο, η αποκέντρωση μερικές φορές οδηγεί σε καταστροφές αν η τοπική διοίκηση, οι τοπικές αρχές δεν χειρίζονται σωστά ε, τα διάφορα θέματα ή τα χειρίζονται υπέρ τους. Οπότε πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ε, και να τις συνοδεύσουμε στην αποκέντρωση. Το Μαρόκο το κάνει πολύ και μας έχει ζητήσει βοήθεια και τη δίνουμε. Ελπίζω λοιπόν ότι και σε αυτό θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Να, το, η μέθοδος αυτή της διδημοποίησης, των αδελφοποίησης, όπως λέγεται, των ε, πόλεων μεταξύ τους, είναι ένας τρόπος για να τις βοηθήσουμε. Λέτε χωρίς ασφάλεια και νομική ασφάλεια κυρίως δεν υπάρχουν ε, επενδύσεις από το εξωτερικό. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό και σε όλες αυτές τις χώρες δουλεύουμε για να βελτιώσουμε την ασφάλεια αυτή στη Λιβύη όπου η κατάσταση είναι πιο δύσκολη, προσπαθούμε να καθιδρήσουμε μία δράση ελέγχου των συνόρων. Στην Τινησία τους προτείναμε εδώ και πάνω από χρόνο να τους βοηθήσουμε να μεταρρυθμίσουν τον τομέα ασφάλειας. Διστάζουν όμως. Και γενικά προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να ενισχύσουν την ασφάλειά τους και να δουλέψουμε και πάνω στο ρυθμιστικό τους πλαίσιο για να ενισχύσουμε τις επενδύσεις. Δεν έχουμε θεαματική επιτυχία, βοηθάμε όμως γιατί ξέρουμε ότι όπως λέτε κι εσείς αυτά αποτελούν μεγάλο εμπόδιο η ανασφάλεια. Τώρα για την ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν μιλάτε στην Τινησία με την κοινή γνώμη, με οργανώσεις για παράδειγμα που εκπροσωπούν γυναίκες, τι σας λένε, σας λένε ότι νιώθουν υποπίεση για το πώς πρέπει να ντύνονται, για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Και πιστεύω ότι σε τομείς, όπως πολύ σωστά είπατε, επί Μπουργκίμπα και Μπεναλή είχαν κατακτήσει κάποια πράγματα, τώρα μας λένε ότι αυτά μπορεί να αμφισβητηθούν υπό την πίεση των σαλαφιστών, για παράδειγμα και είναι οι φίλοι μας και οι συνομιλητές μας στην Τινησία που μας τα λένε αυτά. Αν υπάρχουν τόσο πολλές γυναίκες στην Τινησία που λένε ότι βρίσκονται υποπίεση, ε, προφανώς έτσι θα είναι. Υπάρχει πραγματικά κίνδυνος, δεν τα βγάζουν από το μυαλό τους φαντάζομαι. Κλείνουν για παράδειγμα πάρα πολλέ αίθουσε κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους. Είναι κακό σημάδι να κλείνουν οι κυματογράφοι γιατί νιώθουν ότι απειλούνται. Όπως επίσης η κατανάλωση ποτών. Καλά δεν μιλάω φυσικά για αλκοολισμό, αλλά αν κάποιος θέλει να πιει μια μπύρα και δεν μπορεί να το κάνει, ε, αν δεν είναι γιατρικούς λόγους που το απαγορεύεται, ε, τότε αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Τώρα κατά πόσο πρέπει να ανησυχήσουμε τις γυναίκες, α ναι αυτό σας το απάντησα. Στην Αναγκόμες να απαντήσω τώρα γιατί δυσκολευόμαστε να θέσουμε σε εφαρμογή όλες αυτές τις ωραίες ιδέες. Ένας λόγος είναι πως το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας είναι οι κακές σχέσεις ανάμεσα στην Αλγερία και το Μαρόκο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και αν μέχρι τώρα δεν καταφέραμε να βοηθήσουμε τις χώρες Μαγκρέπ να αναπτύξουν τη συνεργασία μεταξύ τους και την περιφερειακή ολοκλήρωση, είναι κατά κύριο λόγο ακριβώς γι' αυτό. Πώς τώρα να αντιμετωπίσουμε αυτούς που χρηματοδοτούν τους αλαφιστές. Εδώ με φαίνεται σε δύσκολη θέση, γιατί ναι, πράγματι ξέρουμε ποιο τους χρηματοδοτεί, αλλά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε τις καλύτερες σχέσεις του κόσμου μαζί τους. Μπορούμε λοιπόν να θίξουμε πραγματικά και ειλικρινά αυτό το πρόβλημα μαζί τους. Πρέπει να το συζητήσουμε. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβλημα οι χώρες που κατονομάσατε, οι δύο χώρες τις οποίες αναφερθήκατε, επενδύουν πάρα πολύ στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θέλουν να τσακωθούν μαζί τους. Αγοράζουν από την άλλη όπλα. Δίνουν επίσης υλικά τα οποία χρειαζόμαστε, υδρογονάθρακες. Συνεπώς, για ένα σωρό λόγους, είναι προνομιούχη εταίροι των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχετε δίκιο και στη χώρα που γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα τη στιγμή που, να, στη Λιβύη για παράδειγμα, χρηματοδοτούν τους παραστρατιωτικούς. Τους χρειαζόμαστε για άλλους λόγους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τα γεγονότα στην Αλγερία, αν είναι καρπός των εσωτερικών ε, διανέξεων ε, μέσα στην Αλγερία. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοιες ενδείξεις, δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορούμε να κάνουμε ένα σώρο υποθέσεις. Δεν ξέρω όμως. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι στο νότο της Αλγερίας και παρά την επιμονή των Αλγερινών αρχών και, των αποφα... και της αποφασιστικότητάς τους υπάρχουν διάφορες συμμορίες που δρούν και από την Τζιχάτ. και όλα αυτά τα ξέραμε και πριν τις εξελίξεις στο Μαλί και πριν τα γεγονότα στη Λιβύη πριν από δύο χρόνια. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, μερικέ φορέ δεν βλέπουμε μακριά. Παρ' αυτά, πριν από τρία χρόνια είχαμε αρχίσει στρατηγική για την ανάπτυξη και την ασφάλεια στο Σαχέλ. Άρα εδώ και μερικά χρόνια ήδη και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλοι που δρουν στην περιοχή γνωρίζουν ότι στο Σαχέλ υπάρχουν πολλά προβλήματα οργάνωσης ε, εγκληματικών συμμοριών κλπ. Άρα δεν πρέπει να ψάχνουμε στα προβλήματα ε, που έχει στο εσωτερικό της η αλλεργία τα πρόσφατα γεγονότα. Οι ρίζες των όσων έγιναν στην αλλεργία την προηγούμενη εβδομάδα υπάρχουν στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Και βέβαια τα γεγονότα στη Λιβύη πριν από δύο χρόνια και αυτά που έγιναν και γίνονται εδώ και μερικές εβδομάδες στο Μαλί σίγουρα συνεισέφεραν στο να διωγκωθεί το πρόβλημα τι κάνουμε για τη Δυτική Σαχάρα τώρα που κατά πάσα πιθανότητα είναι μία από τις συγκρούσεις που τροφοδοτεί την περιοχή εκεί και τις επιμέρους ε, συγκρούσεις. Η θέση μας ήταν ότι στηρίζουμε τον Κρίστοφερός των Ηνωμένων Εθνών, αλλά γιατί το λέμε αυτό για να είμαστε ειλικρινεί. Γιατί δεν υπάρχει κοινή άποψη μεταξύ των 27. Ορισμένες χώρες στηρίζουν απόλυτα τη θέση του Μαρόκο. Και έχετε και διάφορες χώρες που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να γίνει δημοψήφισμα το οποίο να προσφέρει τη δυνατότητα για ανεξαρτησία στη Δυτική Σαχάρα. Συνεπώ είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε κοινή θέση. Και η απουσία κοινή θέση είναι δύσκολο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δραστηριοποιούνται περισσότερο για το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας. Δεν το δικαιολογώ, σας το εξηγώ αυτό που συμβαίνει. Σας λέω ότι δεν δραστηριοποιούμε θα περισσότερο για αυτό το λόγο. Αυτά, νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ας κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα μέχρι να έρθει η αντιπρόεδρος Κυβέρνησης της Σερβίας. Ciao.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

Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα προβλέπεται ανταλλαγή απόψεων με την Σουζάνα Γκρουμπιεζίκ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της Δημοκρατίας της Σερβίας. Καλωσορίζω την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης που έρχεται για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας Εξωτερικών Υποθέσεων. Τα μέλη της Επιτροπής όμως που επήγαν στη Σερβία και στο Κωσυφοπέδιο είχαν τη χαρά να σε συναντήσουν στο Βελιγράδι. Το 2012 ήταν σημαντική χρονιά για τη Σερβία, διότι έλαβε το καθεστώς της υποψήφιας χώρας και το 2013 είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι είναι το έτος κατά το οποίο η Σερβία θα πρέπει να πληρώσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή μας συζητεί την ετήσια έκθεση πρόοδου για τη Σερβία. Ε, την εξετάσαμε, είναι η έκθεση του κυρίου Κατσίν, σήμερα το πρωί μόλις, και μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ευρεία υποστήριξη ε, στην Επιτροπή υπέρ του έναρξης διαπραγματεύσεων με τη Σερβία, γιατί πιστεύουμε ότι αυτές θα συμβάλλουν έτσι περαιτέρω προς την δημοκρατική ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι ότι ο διάλογος μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας μέσω της ε, Μεσολάβησης της Ένωσης είναι πολύ σημαντικός και φαίνεται ότι επιτελείται καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, στις συνομιλίες. Και οι δύο πλευρές ενδιαφέρονται για την εξομάλυνση των σχέσεων ώστε οι πολίτες της Σερβίας και Κωσοβού να ζήσουν σε ειρήνη και ευημερία. Χωρίς ε, άλλες παρατηρήσεις, σας δίνω το λόγο κυρία Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης για να παρουσιάσετε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Σερβική κυβέρνηση και τους ε, όρους, ε, τις προκλήσεις για τους όρους για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά και τιμή που έχω αυτή την ευκαιρία να απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή εδώ των Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερα αυτή την ενδιαφέρουσα περίοδο όπου συζητείται η πρόοδος της Σερβίας ε, στα θεσμικά όργανα της Ένωσης ε, και συζητείται και το σχέδιο ψηφίσματος στην Επιτροπή σας. Και ως ε, πρώην βουλευτής καταλαβαίνω και εγώ πολύ καλά και εκτιμώ το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην διαδικασία της ολοκλήρωσης των υποψηφίων χωρών όπως η Σερβία. Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων, γι' αυτό δεν θα μακρηγορήσω, θα δώσω ευκαιρία στα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής σας να θέσουν ερωτήσεις και εγώ θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Δεν θα είναι μονόλογος, θα είναι διάλογος αυτός και αυτό το σέβομαι. Στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόοδος της Σερβίας καθοδόν προς την Ευρώπη αναγνωρίστηκε και εκτιμήθηκε και τα συμπεράσματα άνοιξαν τη δυνατότητα της έναρξης ή του ανοίγματο των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον. Αυτό το σχέδιο ψηφίσματος της Επιτροπής της δικής σας επιβεβαιώνει τα ίδια πράγματα και εγκρίνει την, επίσης την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Είναι σημαντικό να οικοδομήσει πάνω σε αυτά τα επιτέγματα η Σερβία και να επιτελέσει πρόοδο σε κύριους τομείς και ζητήματα και να ανοίξουν οι διαπραγματεύσεις ή δυνατόν στο τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας, δηλαδή τέλος Ιουνίου. Ένα πολύ σημαντικός λόγος να πάρουμε ημερομηνία είναι να διατηρήσουμε για να διατηρήσουμε τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων στη Σερβία, ώστε η διαδικασία της ολοκλήρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μια αντιστρέψιμη. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, η μεγαλύτερη πρόκληση ή η βασική πολιτική συνθήκη προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι ο διάλογο με την Πρίστινα. Και χαίρομαι που μπορώ να πω ότι ο διάλογος με την Πρίστινα έχει εδρεωθεί ως μόνιμη αρχή στο Σερβικό Κοινοβούλιο μέσα από το ψήφισμα για το κοσυφοπαίδιο που εγκρίθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Η εξομάλυνση των σχέσεων με την Πρίστινα είναι το ε, εξοκάνευ για την έναρξη ε, Είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα για τη Σερβία, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική καμία στο διάλογο. Εμείς ε, Θεωρούμε ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συνεργαστούν με τρόπο ευέλικτο και ρεαλιστικό, ώστε να καταλήξουν σε δίκαιη και αποδεκτή ε, λύση και να βελτιώσουν τη ζωή των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων στο κοσυφοπαίδιο. Μέχρι τώρα ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων θεμάτων έχουν ε, υπάρξει και ε, ο πολιτικός διάλογος στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο θα συνεχιστεί. Ο τέταρτος γύρος του διαλόγου έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες μόλις, στις 17 Ιανουαρίου, εδώ στις Βρυξέλλες και υπό την αιγίδα της ε, κυρίας Κάθριν Άστον. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναγνωρίσει την πρόοδο στον διάλογο με την Πρίστινα που είναι ορατός, μόνιμος και διατηρήσιμος και βιώσιμος. Η εφαρμογή της συμφωνίας για, το IBM ε, είναι σε πρόοδο και το IBM εφαρμόζεται σε τέσσερα διοικητικά σημεία διέλευσης όπως υποσχεθήκαμε και συμφωνήσαμε. Δηλαδή την ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε και πάντα πρέπει να επιμένουμε στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις στη Σερβία. Η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων συνεχίστηκε μετά το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Συνεχίζουμε να εργαζόμεθα σκληρά ε, δίνοντας μεγάλη προτεραιότητα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, το κράτος δικαίου, τη προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των μειονοτήτων και βεβαίως μεγάλη έμφαση τώρα με την οικονομική κρίση, ε, μεγάλη έμφαση δίνεται στην οικονομία. Η κυβέρνηση ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης με βάση τις συστάσεις και τις προτεραιότητες που αναφέρονται στην έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δημιουργήσαμε ένα εθνικό συντονιστικό φορέα για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος δράσης ε, με επικεφαλή στον Πρωθυπουργό και αυτό έδωσε νέα όφηση στις μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς της ζωής στη Σερβία. Η μεταρρύθμιση του δικαστικού σώματος ή για να είμαι πιο συγκεκριμένη η αντιμετώπιση των ελλειμψέων της προηγούμενης μεταρρύθμισης θα συνεχιστεί να είναι στις προτεραιότητες της κυβέρνησης επίσης. Το πρώτο σημαντικό βήμα ολοκληρώθηκε με βάση την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου οι δικαστές και οι εισαγγελείς επιστρέφουν στην εργασία τους. Η νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, που υπάρχει στο πρόγραμμα δράσης θα υιοθετηθεί όπως μου έμαθα σήμερα μέχρι το τέλος Μαρτίου. Νέα νομοθεσία για τις κρατικές συμβάσεις εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο που ε, αντιμετωπίζει και αποτρέπει ε, καταχρήσεις και επιβάλλει πλήρη έλεγχο της όλης διαδικασίας. Τώρα, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, το νομικό πλαίσιο είναι καλά αναπτυγμένο, τα ανθρώπινα δικαιώματα διασφαλίζονται και προστατεύονται από το Σύνταγμα. Υπάρχει νόμος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μειονοτήτων και υπάρχει και νόμος για την πρόληψη και απαγόρευση συγγνώμη, των διακρίσεων. Όμως ακόμα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για την εφαρμογή των νόμων αυτών. Επίσης να αναφέρω κάποια επιτεύγματα εδώ το Κοινοβούλιο της Σερβίας ε, ολοκλήρωσε το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των ορθών πρακτικών εις ό,τι αφορά τα μέτρα κατά των διακρίσεων. Ε, τώρα 34% των βουλευτών στο Σερβικό Κοινοβούλιο είναι γυναίκες. Κάποια θετικά βήματα έγιναν για να βελτιωθεί η κατάσταση του πληθυσμού των Ρωμά και το ενημερωμένο πρόγραμμα δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής για τη βελτίωση της θέσης των Ρωμά θα τεθεί στην ατζέντα της κυβέρνησης κατά το πρώτο εξάμεινο φέτος. Δουλεύουμε επίσης ε, τη στρατηγική κατά των διακρίσεων ε, και θα έχουμε ένα γενικό έγγραφο το οποίο έχει σχέδιο δραστηριοτήτων για να μειωθεί το επίπεδο διακρίσεων στην κοινωνία μας. Ε, θα εστιάσουμε ε, στην ε, ανάπτυξη ανοχής στις διαφορές, ισότητα, ίσες ευκαιρίες και πρόληψη συγκρούσεων. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στη Σερβία, ε, είναι η έκθεση βιρογνωμόνων της Επιτροπής που εκδόθηκε τον Αύγουστο. Η έκθεση ήταν θετική και δίνει συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Και αυτά όλα τα λαμβάνει η Σερβία πολύ σοβαρά υπόψη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δικαιώματα του πληθυσμού των ΛΟΑΔ, το Σύνταγμα της Σερβικής Δημοκρατίας προστατεύει την αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, ελευθερία γνώμης και έκφρασης, όπως και την ε, ελευθερία του συναθρίζεσαι για όλους τους πολίτες. Ο νόμος κατά των, ε, προ... διακρίσεων προβλέπει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις βάσει του σεξουαλικού προσανατολισμού. Σε εταιρική σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Σερβία συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα που είναι καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το κοινωνικό φύλλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Στις 13 ε, Δεκεμβρίου πέρσι έγινε η πρώτη συνάντηση στο Βελιγράδι για αυτά τα θέματα και αναγνωρίστηκε αυτό στην επιστολή του Επιτρόπου για τη διεύρυνση, στην επιστολή του στα μέλη του Συμβουλίου το Δεκέμβριο. Ο στόχος της διάσκεψης ήταν να υπάρξουν κοινά μέτρα για την εφαρμογή τη σύσταση της Υπουργικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθερότητας και Συνεργασίας, υπάρχει μια ενδιάμεση συμφωνία. Τώρα μπαίνουμε στο πέμπτο έτος της εφαρμογής και στην αρχή του επομένου έτους η Σερβία θα έχει το καθεστώς εμπορική απελευθέρωσης βιομηχανικών και άλλων προϊόντων με εξαίρεση κάποιων στρατηγικής σημασίας προϊόντων. Η εφαρμογή της SAA είναι σημαντική για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ένταξης. Μία προσδοκία που έχουμε είναι ότι το SAA, το, η συμφωνία αυτή σταθεροποίηση και συνεργασία θα, έρθει, θα τεθεί σε εφαρμογή ούτω ώστε η, να κυρώσει και η τελευταία χώρα η Λιθουανία τη συμφωνία μέχρι το, την Άνοιξη. Ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε. Τώρα, η απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πολύ σύντομα να πω δύο λόγια γιατί είναι σημαντικό πολύ για μας αλλά και για την περιοχή των ε, Δυτικών Βαλκανίων γενικότερα. Και θα αναφέρω ορισμένα μέτρα που ελάβαμε για το θέμα αυτό και το πρόβλημα, το πρόβλημα των ψευδών αιτήσεων ε, ασύλου της ε, χώρες μέλη της Ένωσης. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες κάποιες χώρες της Ένωσης για τον αυξημένο αριθμό των ψευδών αιτήσεων ασύλου τους τελευταίους μήνες, αλλά η Σερβία συνεχώς λαμβάνει ε, προληπτικά μέτρα, επικοδομητικά μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα και εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα που μας έχουν συστήσει στην τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την ε, παρακολούθηση του καθεστώτος ε, θεωρήσεων που συζητήθηκε και στο Συμβούλιο Υπουργών στις 25 Οκτωβρίου. Έχουμε ε, τακτική αλλά ανταλλαγή απόψεων και επιστολές ε, έλεγχο των ε, σημείων διέλευσης και παρακολουθούμε τη θέση των μειονοτήτων. Επίσης έχουμε καθορίσει ποινικέ διαδικασίες όταν χρειάζεται ε, και θα διώκονται και θα τιμωρούνται οι ψευδείς ε, τούντες ε, άσυλο. Επίσης έχουμε και νόμο για τη διαχείριση της μετανάστευσης και τους τελευταίους δύο μήνες ο αριθμός των ψευδών αιτήσεων άσυλο σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών μειώθηκε δραστικά συνεπία των μέτρων μας. παράλληλα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η λήψη όλων αυτών των μέτρων σημαίνει ότι πρέπει να ε, είμαστε στα στενά περιθώρια μεταξύ αυστηρών μέτρων και διακρίσεων και η κοινωνία μας δεν θέλει να διακινδυνεύσει επιτεύγματα στα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν αναγνωριστεί άλλωστε στην έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο τελευταίο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολίτες της Σερβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να υποφέρουν από την κατάχρηση ε, του δικαιώματος ασύλου. Έτσι, στη διαδικασία αλλαγή του άρθρου 539, μάλλον 359, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να αλλάξει ο κανονισμός 85 από το 2005. Και με το νέο κανονισμό η Σερβία θα θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα, όπως και η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Ε, έτσι ήταν και εκείνες όταν έγιναν υποψήφιες χώρες το 2005. Επίσης, ε, μεγάλη σημασία αποδίδομαι στην περιφερειακή συνεργασία και όπως βλέπω και στο σχέδιο ψηφίσματός σας και εσείς το αναγνωρίζετε αυτό ως θετικό επίτευγμα της σερβικής κυβέρνησης. Η τελευταία επίσημη επίσκεψη του Κροάτη Πρωθυπουργού στη Σερβία αποδεικνύει έτσι περαιτέρω ότι εμείς προτιθέμεθα και έχουμε δεσμευθεί να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με όλους τους γείτονές μας στην περιοχή. Χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν από την πλευρά μου, ε, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτή την παρέμβαση ευχαριστώντας σας για την προσοχή σας και βεβαίως ε, με χαρά θα ακούσω τις ερωτήσεις σας και τη συζήτηση, τη συμμετάσχω στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Κούκαν, τον πρώτο ομιλητή στον κατάλογό μου, σας θυμίζω ότι σε μισή ώρα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γκίλμορ, Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Το λέω αυτό γιατί σας ζητώ να είστε σύντομοι. Κύριε Κούκαν. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζω πραγματικά από βάθους καρδίας, κυρία Κρούτσπεκ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Σερβίας. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά παρόλα αυτά γνωρίζουμε ότι είσαστε πολύ αφοσιωμένοι στην ατζέντα για την διεύρυνση. Η Σερβία από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση βρίσκεται σε πολύ καλή θετική διάθεση αλλά αυτό σημαίνει ότι έχετε κάποιες υποχρεώσεις απέναντί μας. Δεν μπορεί να μας δημιουργείτε τις ελπίδες ότι είναι στο σωστό δρόμο η Σερβία. Πρέπει να αναλάβετε και την ευθύνη αυτού. Στις αγωγικές σας παρατηρήσεις είπατε ότι υπάρχουν διάφοροι τομείς στους οποίους πρέπει να πετύχετε περισσότερα αποτελέσματα. Χαιρόμαστε που συνεχίζεται ο διάλογος, μιλάμε για την εφαρμογή των τη θέση σε ισχύ δηλαδή των συμφωνιών και σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε όσο πιο υπεύθυνα. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε και θα συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια του διαλόγου σε όλες του τις διαστάσεις. Αλλά πολλά θέματα και αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο εσείς προσεγγίζετε το διάλογο. Η έκθεση και η στάση μας έχει να κάνει και με την αξιολόγηση αλλά και με το τι κάνετε εσείς και τι έχετε πετύχει και τι συνεχίζετε να πετυχαίνετε. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος είναι στην Βρατισλάβα και ότι έκανε μια δήλωση υπέρ της Ευρώπης. Έχει πραγματικά την ικανότητα να μιλάει πολύ ρεαλιστικά για τα διάφορα ζητήματα. Αλλά τελικά το θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι θέμα πάνω στο οποίο από ό,τι φαίνεται δουλεύει η κυβέρνηση της Σερβίας και εμείς σας ανθαρρύνουμε σε αυτό. Έχω μία ερώτηση. Για το περίφημο άρθρο 359. Γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις, ότι είναι στο Κοινοβούλιο ακόμα προσυζήτηση. Πρέπει να ξέρετε ότι εμείς παρατηρούμε από κοντά το τι γίνεται και πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Και θέλω να τονίσω ότι είναι προς το συμφέρον της Σερβίας και ημών βέβαια να μην ακούμε διαμαρτυρίες από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις όπως έγινε στο πρόσφατο παρελθόν. Οπότε η Αντιπρόεδρος θα Ξέρω ότι το γνωρίζει όπως και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μήπως έχετε περισσότερες λεπτομέρειες να μας πείτε δηλαδή πού ακριβώς βρίσκεται η κατάσταση από αυτού σήμερα. Και να προσθέσω ότι θέλουμε πάρα πολύ γρήγορα να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατσίν έχει τώρα το λόγο που είναι εισηγητής για την Σερβία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα αγγλικά όμως. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι η μέρα που βλέπουμε την έκθεση προόδου της Σερβίας και βλέπουμε ότι το γενικό πνεύμα της έκθεσης αυτής είναι θετικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν του σκιώδει ηγητέ που συνέβαλαν στο να καταλήξουμε τελικά σε μια ισοκελισμένη έκθεση η οποία καλωσορίζει τελικά τη Σερβία στις δομές τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω ότι η κυβέρνησή σας κατάφερε μέσα σε μερικούς μήνες να πετύχει πάρα πολλά πράγματα στις σχέσεις με το κοσφοπέδιο. Πρόκειται για ένα πραγματικό επίτευγμα, όχι μόνο για τις σχέσεις με το κοσφοπέδιο, αλλά και για τις σχέσεις σας με τις άλλες χώρες. Αναφερθώ καταρχάς στο Μαυροβούνιο. Ακόμα θυμάμαι τι είχε πει τότε ο Πρωθυπουργό Κοστούνιτσα ότι δεν επρόκειτο ποτέ να αναγνωρίσουμε την ανεξαρτησία του Μαυροβονίου, πράγμα το οποίο το κάνανε στη συνέχεια. Τώρα όμως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ θετικό παράδειγμα για όλες τις όμορές σας χώρες. Τα όσα υπόθηκαν κατά την επίσκεψή σας στη Βοσνία ήταν πάρα πολύ θετικά για όλους εμάς. Όσον αφορά τώρα τον διάλογο με το κοσφοπέδιο, αυτό το οποίο θέλω να υπογραμμίσω το ακόλουθο. Εγώ θα ήθελα όχι μια επιτυχία μόνο στον 6ο και 7ο διάλογο, αλλά επιτυχία στον 8ο, 9ο, 10ο και ούτω καθεξής. Ο Απρίλιος 8 ο το ο 10 ο και το καθεξης ο απριλιος ειναι οντω η καταληκτική μας ημερομηνία, θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν όλες αυτές οι ημερομηνίες που έχουμε για να καταφέρουμε να πετύχουμε καλύτερη σχέση με το κοσφοπέδιο, όσον αφορά την καταπολέμηση της συστημικής διαφθοράς και του εγκλήματος. Πρέπει όντω να αναγνωρίσω ότι έχετε κάνει πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Από την άλλη όμω, τα πράγματα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Βλέπουμε ότι ο κίτρινο τύπο έχει όλε αυτέ τι λεπτομέρειε εκ των προτέρων μάλιστα, για όλε τι έρευνε, οι οποίε γίνονται. Δεν είναι δημοκρατικά πρότυπα αυτά. Γίνονται εκ των προτέρων ανακοινώσεις, δίδονται πολύ συγκεκριμένε λεπτομέρειε, εκ των προτέρων διαραίουν στον κίτρινο τύπο όσον αφορά την έρευνα εγκλημάτων και διαφθοράς. Πραγματικά αυτό είναι επέσχυντο και πρέπει να κάνετε κάτι προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Δεν θα ήθελα να αφαιρθώ στο άρθρο 359. Οι συνάδελφοί μου άλλωστε θα πούνε πολλά περισσότερα πράγματα από αυτού. Αυτό που θέλω να πω είναι το ακόλουθο. Οτιδήποτε και να κάνετε, παρακαλώ πολύ, μην κάνετε κάτι για μας. Οτιδήποτε και να κάνετε, κάντε το για τους δικούς σας τους πολίτες, για την εμπιστοσύνη που αυτοί θα πρέπει να έχουν προς την κυβέρνησή σας, για το γενικότερο ευρωπαϊκό πνεύμα και για ένα καλύτερο μέλλον για τη νέα γενιά της Σερβίας που προσβλέπει σε εσά και περιμένει και νέες θέσεις εργασίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε ο κύριος Πόσελτ για δύο λεπτά. Κύριε Αντιπρόεδρε, είμαι υπέρ της ε, ένταξης της Σερβίας. Επίσης την προσωπική σας εργασία την θαυμάζω, όπως και το έργο του κόμματό σας. Όμως θα κάνω δύο πολύ επικριτικ... Ε, ε, κρίσιμες ερωτήσεις. Πρώτον, το καθεστώς του κοσυφοπεδίου που συζητείτε συχνά. Εγώ χαιρετίζω τις συνομιλίες και τις πρακτικές διευκολύνσεις, αλλά Διαρκώς στη χώρα σας υπάρχουν φωνές που θέτουν το θέμα του καθεστώτος. Επειδή οι γυναίκες είναι πιο θαραλέες συνήθως από τους άνδρες, πρέπει να σας πω ότι οι Σέρβοι πολιτικοί θα πρέπει να έχουν το θάρρος να πούν στο λαό τους κάποια στιγμή ότι το Κόσοβο δεν θα ξαναγίνει σερβικό. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει σχέση καλής γειτονία και η ολοκλήρωση της Σερβίας είναι το μέλλον στην Ένωση. Ε, δεύτερον, Έχουμε την οξία κρίση στον Πρέσεβο. Ξέρω την περιοχή πολύ καλά. Έχω πάει συχνά εκεί. Παρακαλώ να κάνετε το παν για να ελαφρύνετε την έσχατη ένδια εκεί, ε, τα σοβαρά προβλήματα, τα προβλήματα ε, επικοινωνίας με το Κωσυφοπέδιο και τη Μακεδονία μέσα από περιφερειακά σημεία διέλευσης αν δεν τονωθεί η οικονομία στην περιοχή αυτή θα γίνει εστία κρίσης για το μέλλον, στο μέλλον. Παρακαλώ λοιπόν να φροντίσετε ιδιαίτερα για την περιοχή αυτή. Θαυμάσια κύριε Πόστηλε. Η κυρία Γκόμες, δύο λεπτά. Κύριε Υπουργέ, είμαστε πολύ υπέρ της έναρξης των διαπραγματεύσεων με τη Σερβία φέτος. Όπως ξέρετε και το είπατε και ίδια, οι σχέσεις Βελιγραδίου Μελιγραβίου-Πρέστινας είναι πολύ σημαντικές και θέλω με συνεργασία με την Γιούλεξ από την πλευρά σας και αυτή την ερευνητική ομάδα, ε, την Task Force και θα πρέπει να υπάρξει στο βόρειο τμήμα της χώρας αποφυγή διπλών αστυνομιών και δικαστικών σωμάτων. Εμείς ετοιμάσαμε, αν θέλετε, το δρόμο για το διάλογο. Εσείς μπορείτε να μας πείτε αν το πιστεύετε αυτό και ε, αυτό έχει γίνει κατανοητό από τον κόσμο από τις δύο πλευρές. Για τις μεταρρυθμίσεις για το κράτος δικαίου. Ο κύριος Κατσίν ανέφερε τις ε, ανησυχητικές εξελίξεις ε, με τα άρθρα στον τύπο που είναι τελείως αντιφατικά στην καταπολέμηση του διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος βέβαια θέλουμε οπωσδήποτε πρόοδο και τα μέσα ενημέρωσης έχουν κεντρικό ρόλο εδώ τα οποία αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προσκόμματα στην ελεύθερη λειτουργία τους στην Σερβία. Τι σχεδιάζετε να κάνετε για να αντιμετωπίσετε το θέμα έλλειψης διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης στη Σερβία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Λούνατσεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα εξ ονόματος της ομάδας των Πρασίνων να καλωσορίσω την Αντιπρόεδρο και χαίρομαι που την βλέπω ξανά μετά τη συνάντησή μας στο Βελιγράδι. Καλώς ήρθατε. Συνεχίζω αυτά που είπε ο κύριος Κατσίν στο τέλος της παρέμβασής του. Ε, αυτά που πρέπει να κάνετε για τους πολίτες σας, ε, για ένα ευρωπαϊκό πνεύμα στη χώρα. Εμείς ε, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί όταν ήρθε η κυβέρνηση και εγώ. Πρέπει να πω ότι είδαμε όμως ότι μετά αλλάξαμε γνώμη γιατί βελτιωνόταν τα πράγματα. Ε, θέλουμε ακόμα καλύτερα να πάνε τα πράγματα. Τώρα για ένα θέμα. Είπατε πόσο σημαντικό θεωρείτε το θέμα των ίσων δικαιωμάτων και μη διακρίσεων των ΛΟΑΔ, δηλαδή λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αμφιφίλων. Ε, υπάρξει, υπάρχει πρόοδος. Δεν είδαμε ε, το, ε, ακόμα την ε, παρέλαση, ε, αλλά... Υπήρξαν στοιχεία hooligans, τα οποία δεν ε, πήγαν στη δικαιοσύνη, δεν προσήχθησαν στη δικαιοσύνη, γιατί ε, υπήρχαν ε, από προηγούμενες παρελάσεις προβλήματα. Θα πρέπει να φροντίσετε για την ασφάλεια. Ε, εγώ είμαι εισηγήτρια για το κοσυφοπαίδιο και συζητήθηκε το θέμα σήμερα. Η ψηφοφορία θα γίνει σε δύο εβδομάδες. Εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που είπατε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στο διάλογο. Και όπως προείπα, σημειώθηκε πρόοδος άνευ προηγουμένου πρόοδος όπως στην ολοκληρωμένη διαχείριση συνόρων. Ε, προβλέπεται ότι θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ των Προέδρων Νίκο, Νίκολης και Γιαγιάγκα. Ε, υπάρχει ημερομηνία και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε γιατί τα ακούσαμε μένα αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία. Ε, κάτι που συζητείται στο διάλογο αλλά χωρίς αποτελέσματα και είναι η τελευταία μου πρόταση κύριε Πρόεδρε παράλληλες δομές στο βόρειο κοσυφοπέδιο. Ε, θα καταργηθούν στο, στην αστυνομία και στο δικαστικό σώμα και θα υπάρχει επίσης μία διαφανή σχέση και σε θέματα υγείας και παιδείας με την κυβέρνηση της Πρίστινας. Ο κύριος Τάνοκ, δύο λεπτά. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε σας καλωσορίζω εξ ονόματος της ομάδας ECR. Θεωρούμε ότι η Σερβία είναι φίλη χώρα. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη χώρα σας. Είδαμε και την έκθεση για τη Σερβία σήμερα και καλωσορίζουμε βέβαια τις μεταρρυθμίσεις που κάνετε για μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότερη δημοκρατία, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον άκουσα τα όσα είπατε για τα δικαιώματα λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αμφιφιλόφιλων και διεμφυλικών. Θα ήθελα να αναφερθώ καταρχάς στο άρθρο 359. Πολλοί Σέρβι Πίκοι από τη δική μου εκλογική περιφέρεια στο Λονδίνο μου λένε ότι χρησιμοποιείται καταχρηστικά το άρθρο αυτό και κατά αυτόν τον τρόπο α, εσείς χρησιμοποιείτε ή καταχράσουσαστικά τη δική του στην περιουσία. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω τι θα κάνετε με το άρθρο αυτό το οποίο έχει παραμείνει ουσιαστικά από το κομμουνιστικό Ιουκοσλαβικό καθεστώς. Επίσης η ομάδα μου είναι υπέρ του διαλόγου Βελιγραδίου Πριστίνας. Υποστηρίζουμε την έννοια ανταλλαγής εδαφών για ειρήνη. Βλέπουμε επίσης όμως ότι υπάρχουν κάποιες εντάσεις στο Πρέσεβο και αυτό μας δημιουργεί ανησυχίες. Γίνανε και κάποιες δηλώσεις για μια μεγαλύτερη Αλβανία. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα σύνορα δυστυχώς δεν είναι ακόμα παγιωμένα στην ε, περιοχή σας και θέλουμε να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον με το ζήτημα του κοσφοπεδίου ή αν τελικά οδηγηθούμε στη μόνη λύση, δηλαδή σε μια διάσπαση του κοσφοπεδίου. Θα ήθελα να συγχαρώ για τις βελτιωμένες σχέσεις με το Μαυροβούνιο, είμαι εισηγητής για το Μαυροβούνιο και είμαι υπέρ της πρόσφατης επίσκεψής σας στην Ποτκορίτσα και για τις επαφές που έχει η κυβέρνησή σας με την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου, καθώς επίσης και με την συμφωνία εκείνη που επιτρέπει την δικαστική εκδίωξη των εγκληματιών πολέμου οι οποίοι είχαν βρεθεί, είχαν βρεθεί στον Μαυροβούνιο. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρετε γρήγορα να προχωρήσετε στι ταξιακέ διαπραγματεύσει. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Κυρία Αντιπρόεδρε τη Κυβέρνηση, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας, για τις παρατηρήσεις σας, για όλο αυτό το ενδιαφέρον το οποίο δείχνετε για τη Σερβία. Σα ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, ο κύριο Ρούτσαρτ, να πάρω το λόγο. Κύρια Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εξ ονόμετος των Σοσιαλιστών και Δημοκράτων πρέπει να σας πω ότι είμαστε σαφώς υπέρ της προσχώρησης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει προφανώς να επιτελέσετε κάποια πρόοδο, αλλά μπορείτε να στηρίζεστε στη δική μας την υποστήριξη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιβραβευθεί για τις μεταρρυθμίσεις της η Σερβία και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Αυτό που θα ήθελα να πω μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που ακούστηκαν είναι το ακόλουθο θα μπορούσε να μα πείτε κάποια πράγματα για τι οικονομικέ μεταρρυθμίσει. Γιατί αλήθεια είναι ότι εμεί εστιαζόμαστε περισσότερο στι πολιτικέ μεταρρυθμίσει στη σχέση με τι γειτονικέ σα χώρε, αλλά ξέρουμε ότι και ο λαό τη Σερβία πέρασε πολύ δύσκολου καιρού τα τελευταία 20 χρόνια. και Υπάρχουν πολλοί που δεν βλέπουν τελικά ακόμα το φω στο βάθο του τούνελ. Τι μπορείτε λοιπόν να μα πείτε, τι μπορεί να κάνει η Σερβία από οικονομική πλευρά και πώ μπορούμε να βοηθήσουμε στα πλαίσια της ενταξιακής διαπραγμάτευσης στους ανθρώπους της Σερβίας, πώς μπορούμε να δώσουμε νέα όθηση στην οικονομία σας, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την οικονομική ανάπτυξη, πώς μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία. Τα όσα είπε ο κύριος τα αληθεύουν όχι μόνο στην περιοχή του Πρέσερο αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές Σερβίας υπάρχουν άνθρωποι που πλήττονται από την ένδια και πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, ποιε είναι οι οικονομικέ μεταρρυθμίσει που προωθείτε. Ευχαριστώ. Και για άλλη μια φορά σα το συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ για τι παρεμβάσει σα. Πάντα μ' αρέσει να μιλάω για την οικονομία, αλλά θα αρχίσω από την αρχή. Πολλοί ευρωβουλευτέ ρώτησαν για το άρθρο 359. Μια αλλαγή δηλαδή στο ποινικό δίκαιο. Βρίσκεται στο Κοινοβούλιο αυτή την εποχή. Δεν έχει ακόμα ψηφιστεί και θα σας εξηγήσω κάπως σύντομα ποια είναι η αλλαγή που προβλέπετε. Αλλά δεν μπορώ να σας πω πότε ακριβώς θα υιοθετηθεί και ποια θα είναι η τελική μορφή του άρθρου. Η πρόθεση είναι να μειωθεί η πίεση που δέχονται οι ιδιοκτήτες επί του παρόντος και πώς δηλαδή να αντιληφθούμε την κατάχρηση ε, σε βάρος ε, της επιχείρησης. Το άρθρο 359 με διαφορετικό βέβαια τρόπο, θα παραμείνει στο ποινικό δίκαιο. Γιατί προς το παρόν υπάρχουν 4.000 υποθέσεις στη δικαιοσύνη που βασίζονται στο άρθρο αυτό. Θα υπάρξει δηλαδή αλλαγή, αλλά δεν θα διαγραφεί από τον ποινικό κώδικα, από το ποινικό δίκαιο. Και αυτό γιατί οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο ανεξάρτητοι και αν είναι, μπορούν να ζημιώσουν ε, μικρούς ε, μετόχους. Συνεπώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσπαθεί να βρει μια ισορροπία ανάμεσα, όπως είπε και ένας ε, ευρωβουλευτής, στην κληρονομιά που έχουμε από το παλιό κομμουνιστικό καθεστώς και τη σημερινή κατάσταση. Πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι υπέρ βεβαίως του κράτους δικαίου και τον, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία. Αλλά ε, δεν έχει συζητηθεί ακόμα, όπως σας είπα, στο Κοινοβούλιο η αλλαγή αυτή, οπότε δεν μπορώ να προκαταλάβω την τελική μορφή του άρθρου. Αργότερα, όταν θα έχει υιοθετηθεί, θα μπορώ να σας πω με ποια ακριβώς μορφή θα συμπεριληφθεί και στο ποινικό δίκαιο. Κάποιοι ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν επίσης στα γεγονότα στην κοιλάδα του Πρέσεβο και με το μνημείο και τι έγινε με την μειονότητα των ε, Αλβανών. Στο κέντρο του Πρέσεβο είχαμε το μνημείο, το οποίο είναι αφιερωμένο ε, στο τι έγινε όταν προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε την ε, τρομοκρατία. Εμείς σαν υπεύθυνη χώρα Είχαμε τρει εβδομάδε διάλογο με τους εκπροσώπους της Μιανότητας των Αλβανών και συμμετείχαμε και στο διάλογο της ΟΕΣΕ και με μέλη της διεθνού κοινότητας. Είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της Σερβίας και δεν υπάρχει κανένα λόγος να επηρεάζει τα πράγματα στην περιοχή. Είναι ένα μήνυμα στο κέντρο του Πρίσεβο που φτιάξαμε το, σε σχέση με την τρομοκρατία το 2001. Πάντως, εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο και ο διάλογος με τους εκπροσώπους της αλβανικής μειονότητας θα συνεχιστεί, ώστε τέτοιου είδους επεισόδια να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Και ως ε, απάντηση ήταν ότι συλλητήθηκαν διάφοροι τάφοι στο κοσυφοπέδιο. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή απάντηση, για να το πω δηλαδή έτσι κάπως ευγενικά. Από τη μια δηλαδή έχουμε το μνημείο, από την άλλη μεριά έχουμε τους ευρικούς τάφους. Με τον κύριο Πάσεκ πάντως ε, έχουμε πει ότι πρόκειται για μια φτωχή περιοχή ε, αλβανική, ότι χρειάζονται πολλές επενδύσεις και μεγάλη βοήθεια από τη χώρα και από επενδυτές, έτσι ώστε η φτώχεια, η ανεργία και όλα αυτά τα αρνητικά αισθήματα που υπάρχουν σε αυτό το μέρος της κεντρικής ε, Σερβίας να απαλληφθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι μια δικασία δηλαδή που προχωράει. Είμαστε όμως σε συνεχή διάλογο, όπως σας είπα, με εκπροσώπους της αλβανικής μειονότητας στη Νότια Σερβία και στο Πρέσοβο. Όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και τι διαβάζουμε στα μέσα ενημέρωσης για συλλήψεις κλπ. Πρόκειται για μερικές μόνο εφημερίδες που γιατί ο τύπος βασικά θέλουμε να εφαρμόσει και να ε, συμμορφωθεί προς τους νόμους που έχουμε ψηφίσει και έτσι ως πολίτες της Σερβίας να γνωρίζουμε ποιοι βρίσκονται από πίσω και ποιος είναι υπεύθυνο αν γίνεται κατάχρηση πληροφοριών από την αστυνομία ή από τη δικαιοσύνη και εμφανίζονται σε αυτές τις εφημερίδες, τα tabloids. Δουλεύουμε πάντως για να τεθούν σε εφαρμογή οι νόμοι που έχουν να κάνουν με τη στρατηγική απέναντι στον τύπο. Δυστυχώ, φτάσαμε στο 2011 για να έχουμε την νομοθεσία αυτή. Αν είχαμε έτοιμη την νομοθεσία νωρίτερα θα είχε λυθεί το πρόβλημα τουλάχιστον μερικώ ω σήμερα. Όσον αφορά τώρα τη συνάντηση του πρόεδρου Νίκολίτ με τον Χάργα, εγώ δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι η ημερομηνία. Ξέρω ότι υπάρχει πρόθεση και υπάρχει το μήνυμα ότι θα γίνει η συνάντηση αυτή. Αλλά πόσο γνωρίζω δεν ξέρουμε πότε. Ελπίζουμε σύντομα. Γιατί όπως είπα και πριν, ο διάλογος είναι μόνιμος βάσει κοινοβουλευτικής απόφασης, οπότε η συνάντηση μεταξύ των δύο θα συνεισφέρει στην ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό μας και τον Πρωθυπουργό του Κωσυφοπεδίου. Με ρωτήσατε επίσης για παράλληλους ε, θεσμούς στο Βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί μεταξύ των δύο και είμαι σίγουρη ότι μέσα από το διάλογο θα καταλήξουμε σε αποδεκτές και για τους δύο λύσεις. Γιατί αυτό που υπερισχύει είναι ότι οι παράλληλοι θεσμοί είναι θεσμοί που υπάρχουν μόνο στο Κωσυφοπαίδιο. Εμείς θέλουμε να λυθεί το ζήτημα πάντως με τις αρχές του Κωσυφοπεδίου και με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η δικιά μας τουλάχιστον πρόθεση. Σύντομα τώρα να αναφερθώ στην οικονομία γιατί ξέρω ότι μιλάω πολύ. Λοιπόν, η οικονομία είναι ένα σημαντικό θέμα. Η Σερβία είναι μια χώρα που προσπαθεί να βγει από την οικονομική κρίση. Η νέα κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μέτρα όχι τόσο φιλολαϊκά, αλλά προκειμένου αν μη τι άλλο να μειώσει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Εγκρίθηκε ο νέος προπολογισμό τον Οκτώβριο που μας πέρασε και το έλλειμμα από 7 θα πάει στο 3,5%. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ την μακροοικονομική σταθερότητα στη Σερβία. Η νέα κυβέρνηση επίσης αναγκάστηκε να αυξήσει κατά 2% το ΦΠΑ, αλλά το 20% είναι ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ΦΠΑ στην περιοχή. Δεν χρειάζεται να πάρουμε μέτρα μείωσης μισθών και συντάξεων. Έχουν όμως παγώσει όσον αφορά την ονομαστική αξία. 2% θα είναι η αύξηση το πολύ. Όσον αφορά τώρα νέες επενδύσεις, για να μειωθεί η ανεργία, θα χρησιμοποιήσουμε τις επενδύσεις αυτής, ανεργία η οποία είναι υψηλή ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Η συνέπεια είναι ότι βλέπουμε να φεύγουν πολύ δυνατά μυαλά από τη χώρα, και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Καναδά, γιατί εκεί μπορούν πιο εύκολα να βρουν δουλειά από ό,τι στη Σερβία σήμερα. Η Παγκόσμια Τράπεζα όμως, το Εθνές Ομοσπονδιακό Τεμείο κλπ. προβλέπουν 2% ανάπτυξη για φέτος στη Σερβία. Αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα θα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσωπικά εγώ όμως δεν πιστεύω ότι θα καταλάβει ε, την θετική αυτή κατάσταση ο κόσμος ε, φέτος. Θα πάρει κάποιο χρόνο παρά τις επενδύσεις που φτάνουν στη Σερβία, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από αλλού. Ε, φυσικά είμαστε και αποδέχτες της προενταξιακής αρρωγής. 200 δις το χρόνο, είπε χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά 90% που είναι το πιο μεγάλο ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες που ήταν στην ίδια κατάσταση που σημαίνει ότι η δίκησή μας είναι έτοιμη να απορροφήσει τα κονδύλια υπέρ των πολιτών της Σερβίας. Αν τώρα κάτι ξέχασα, παρακαλώ να μου το επενθυμίσετε. Ανέ ναι, για τα δικαιώματα των ε, ε, μειονοτήτων και τα δικαιώματα των ομοφιλόφιλων ε, κλπ. Εγώ πιστεύω ότι τελικά την παρέλαση αυτή θα την έχουμε φέτος και ότι οι εξτρεμιστικές ομάδες δεν θα μας εμποδίσουν. Πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτή είναι η πεποίθησή μου, γιατί η κυβέρνηση κάνει τα πάντα προκειμένου να διευκολύνει την κατάσταση όσον αφορά τον ε, πληθυσμό αυτών, τον ε, ΛΑΕΔ, και έτσι πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει εμπόδιο και θα λάβει χώρα φέτος η παρέλαση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι. Πέντε λεπτά διάλειμμα.

Kolleginnen Kollegen, darf ich Sie... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ πολύ ώστε να ξεκινήσουμε. Τελευταίο σημείο στη ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω στην Επιτροπή μας τον Ιρλανδό Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου, τον κύριο Έαμον Γκίλμορ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Ιρλανδικής Προεδρίας και προφανώς θα ασχοληθεί με τα ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων στο Συμβούλιο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας Ξέρω ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με το ζήτημα τη διεύρυνση Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα για την Ιρλανδική Προεδρία. Εμεί σήμερα εξετάσαμε πολλέ εκθέσει πρόοδου στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή για την Κροατία, τη Σερβία και άλλε χώρε και τι επόμενε εβδομάδε θα ψηφίσουμε αυτέ τι εκθέσει. Και ξέρουμε ότι η προσχώρηση των κρατών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντική. Και πρέπει να δούμε βέβαια αν μπορεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση να απορροφήσει τις χώρες αυτές σε μια περίοδο κρίσης. Αυτό που έχουμε δει όμως γενικά είναι ότι με την γενικότερη υποστήριξη και συνεργασία μπορούμε να ξεπεράσουμε ακόμα και την κρίση. Αυτό το είδαμε έμπρακτα και στη δική σας τη χώρα. Και τα όσα έχετε πράξει στην Ιρλανδία θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση και για τους υπόλοιπους. Ξέρουμε ότι η πολιτική γειτονίας και η πολιτική που έχει να κάνει με την Νότια Ευρώπη περνάει από μια δύσκολη φάση και γνωρίζουμε ότι θα υπάρχουν και διαπραγματεύσεις όσον αφορά τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις που θα μας έρθουν από το Συμβούλιο θα μας επιτρέψουν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε γρήγορα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Θα συμπεριλάβουμε και τη λογοδοσία, απόδοση ευθυνών, η Ιρλανδία που έχει παράδοση στο θέμα αυτό θα λάβει τις σωστές αποφάσεις παρά τις πιέσεις που θα προέλθουν από κάποιες ε, χώρες μέλη. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα εργασίας που θα μας βοηθήσει στο μέλλον. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Thank you uh, very much, Mr. Um, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνεται η ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο στην Επιτροπή ΑΦΕΤ Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω ευθύς εξ αρχής να πω ότι και ε, ε, εγώ προσωπικά και η Ιρλανδία εκτιμούμε ιδιαίτερα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ιδιαίτερα στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων. Είχα το προνόμιο να σας συναντήσω κύριε Πρόεδρε πριν από λίγους μήνες και τότε συζητήσαμε την προσέγγιση που θα υιοθετούσε η Ιρλανδική Προεδρία στα διάφορα θέματα και μου καταστήσατε σαφέστατο πρέπει να πω, σαφέστατη την επιθυμία σας να με δείτε το ταχύτερο δυνατό τον Ιανουάριο. Να με λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να έρθω. Ναι, δείχνετε, ε, φοράτε τα, τα εθνικά χρώματα. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εγώ δεν έχω την πολυτέλεια σε καιρούς λιτότητας. Και θα πρέπει μία να κρατήσει έξι μήνες δεν μπορεί να φοριέται καθημερινά λοιπόν, να μην χαλάσει. Ξέρω ότι επί δύο ημέρες συζητείται εντατικά τα θέματα της διεύρυνσης και εξετάζετε την, ε, τις εκθέσεις πρόοδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σειρά χωρών. Ότι είχατε συζήτηση με την Σέρβα Υπουργό Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ξέρω πόσο υποστηρικτική είναι η Επιτροπή σας σχετικά με τα γενικά θέματα και στόχους της πολιτικής διεύρυνσης. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι είναι πρέπον να έρθω στο τέλος αυτής της μακράς συνεδρίας για να συζητήσουμε τις προτεραιότητες για τη διεύρυνση της Ιρλανδικής Προεδρίας. Ε, προσβλέπω να συνεργαστώ στενά μαζί σας για να προχωρήσει η ατζέντα της διεύρυνσης κατά την Προεδρία μας. Θα επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου στην ατζέντα της διεύρυνσης στους επόμενους μήνες. Παράλληλα όμως έχω επίγνωση της νομοθετικής ατζέντα που ε, αφορά την Επιτροπή σας ιδιαίτερα τις προτάσεις για τα εξωτερικά μέσα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας διαβεβαιώνω ότι προσβλέπουμε στην συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας πάνω σε αυτά τα θέματα επί Προεδρίας μας. Πριν μπω στι λεπτομέρειες, ε, επιτρέψτε μου ορισμένα σχόλια σχετικά με τις συνολικές προτεραιότητε Προεδρία τη Ιρλανδίας και πώς αυτές συμπληρώνουν την πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε βεβαίω ότι το σύνθημα της Προεδρίας μας είναι σταθερότητα θέση εργασία και ανάπτυξη. Η Ιρλανδική Προεδρία θα είναι μια Προεδρία χώρα ανάκαμψη που θα προωθεί την ανάκαμψη στην Ευρώπη. Το επίσημο πρόγραμμα της Προεδρίας μας παρουσιάζει λεπτομερώς νομοθετικές και άλλες προτεραιότητες σε όλους τους σχηματισμούς των Συμβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές προτεραιότητες συνοψίζονται ως εξής. Διασφάλιση της σταθερότητας, επένδυση σε ε, διατηρήσιμες θέσεις εργασίας ε, και ανάπτυξη βιώσιμη. Η Ευρώπη και ο κόσμος, ιδιαίτερα τη σημασία του να βλέπουμε πέρα από τα σύνορά μας και να ε, έχουμε σχέσεις με παγκόσμιους εταίρους. Σε σχέση με αυτό το τελευταίο θα συνεργαστούμε στενά με την ύπατη εκπρόσωπο, Πρόεδρο Κάθριν Άστον και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να αντιμετωπίσουμε ε, προκλήσεις κλειδιά στην εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια. Προσβλέπω επίσης το να συνεργαστώ με την Επιτροπή σας, ε, ε, υποστηρίζοντα την ε, είπατε εκπρόσωπο στην Προεδρία μας. Είναι σημαντική θέμα κλειδί η διεύρυνση στην Προεδρία. Η πολιτική διεύρυνση είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο της Ένωσης, στηρίζοντας τη μεταρρύθμιση και το μετασχηματισμό στην Ευρώπη. Η ε, έγκριση και η υιοθέτηση από τα Δυτικά Βαλκάνια και άλλες χώρες υποψήφιες των αξιών της Ένωσης διασφαλίζει τη σταθερότητα και μια αντιστρέψιμη πολιτική μεταρρύθμιση. Είναι προφανή οικονομικά ωφέλη με την ε, μορφή μεγαλύτερη κοινή αγορά που μεταφράζεται σε θέσει εργασία, οικονομική ανάπτυξη και για την Ένωση και τα νέα μέλη. Σε τελευταία ανάλυση η πολιτική αυτή συμβάλλει και στην ασφάλεια και στην ευημερία μα. Η Ιρλανδία από πρώτο χέρι ευίωσε αυτέ τι θετικέ επιπτώσει. Τώρα έχουμε την 40η επέτειο από την προσχώρηση της Ένωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε. Η συμμετοχή ήταν κινητήρια δύναμη για πολιτική τη Ένωση στην Ένωση που ήταν μία από τις τρεις χώρες προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Την τελευταία μας προεδρία του 2004 καλωσορίσαμε 10 νέα κράτη-μέλη. Ε, το 2013 η Ιρλανδική Προεδρία θα συνεχίσει να θέτει προτεραιότητες ε, να θεωρεί προτεραιότητα μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνση πάνω στην, ε, αρχή τη αιρεσιμότητα. Συζητάμε τη διεύρυνση, είναι σημαντικό όμω να βλέπουμε και τη γενικότερη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, η πιο πετυχημένη στις φιλελληνικές διαδικασίες παγκοσμίω. Η πολιτική διεύρυνση είναι από τι πιο επιτυχημένε πολιτικέ γιατί συμβάλλει στα γενικότερα θέματα και τι φιλοδοξίε τη Ένωση. Το όραμα του Ρομπέρ Σουμάν ήταν ένα, μια υπερεθνικής που θα συμμεριζόταν στρατηγικούς πόρους όχι μόνο για να κάνει τον πόλεμο αδιανόητο αλλά και ουσιαστικά και υλικά αδύνατο ε, ούτως ώστε να έχει διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη. Ε, αυτά τα επιτεύγματα ε, ε, εδρεώθηκαν και με το Νομπέλ που δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Άλφρεντ Νόμπελ ε, ήθελε να πηγαίνει το βραβείο σε αυτούς που έκαναν την καλύτερη δουλειά για την αδερφότητα των, των λαών. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα δημιούργησε επίπεδο συνεργασίας, αν προηγουμένου μεταξύ των χωρών αυτή η συνεργασία επέτρεψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει η πιο επιτυχής δύναμη εκδημοκρατισμού και ειρήνης στον κόσμο σήμερα. Η διεύρυνση είναι κεντρική σημασία ε, σε αυτό το επίτευγμα. Η Ιρλανδία πάντοτε ήταν και εξακολουθεί να είναι ε, ισχυρό υπέρμαχο τη διεύρυνσης, Ένωση και του ευρωπαϊκού μέλλοντος των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλουμε συγκεκριμένη πρόοδο στη διαδικασία προσχώρηση για όλε τι υποψήφιε και μελλοντικέ υποψήφιε χώρε. Με αυτή την ευκαιρία πρέπει να αποτίσω φόρο τιμή στον κεντρικό ρόλο που έπεσε το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σα για τη διεύρυνση τη Ένωση. Εσείς είστε, ε, κάθε μεμονωμένο μέλος παίζει σημαντικό ρόλο, διότι μεταφέρει μηνύματα για τι αξίε τη Ένωση στα υποψήφια κράτη-μέλη. Ε, ε, νομίζω ότι στους στόχους μας συμφωνούμε απολύτως με το Κοινοβούλιο. Γενικά το 2013 θα έχει πολλές εκδηλώσεις και θα γίνουν πολλά στη διεύρυνση. Τα τελευταία χρόνια η Προεδρία του πρώτη του εξαμήνου ε, δεν είχε πάρα πολύ δουλειά στο Συμβούλιο ως διεύρυνση. Η Δανεινική Προεδρία τα άλλαξε αυτά με το αποφάσεις που έλαβε για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου προβλέπουν την δυνατότητα να ληφθούν παρομοίως ε, σημαντικές αποφάσεις για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία, το Κουσυφοπαίδιο και ενδεχομένως και την Αλβανία επί Ιρλανδικής Προεδρίας. Και βεβαίως θα δούμε την ολοκλήρωση του ταξιδιού της Κροατίας προς την ε, ένταξη ε, την 1η Ιουλίου. Η δυναμική από την ε, προσχώρηση της Κροατίας θα πρέπει να διατηρηθεί. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων είναι μη αμφίσιμη, αλλά θα πρέπει να παραμείνει και πιστευτή. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου συμφώνησαν αριθμό παραγράφων ραντεβού που προτείνουν να επιστρέψουμε στο πρώτο μισό του 2013 στη δυνατότητα έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξη για τη ΣΟΕΡΔΙΑ και την πρώην Κωνσταντική Δημοκρατία της Μακεδονίας ε, να χορηγηθεί καθεστώ υποψήφια χώρα στην Αλβανία και να ανοίξουν οι διαπραγματεύσει για τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση με το Κωσυφοπαίδιο. Οι αποφάσει επί αυτών των θεμάτων θα ακολουθήσουν από εκθέσει που θα υποβληθούν στο Συμβούλιο των, την Άνοιξη και θα εξαρτηθούν και από τις πρόοδους που θα επιτευχθούν από, την κάθε χώρα. Η Ιρλανδική Προεδρία θα ε, είναι επικεφαλής στην αξιολόγηση του Συμβουλίου. Θα είναι μια λεπτή ισορροπία να δώσουμε χρόνο για να υπάρξει πρόοδος ε, και να αναφερθεί αυτή, ενώ θα διασφαλίζουμε ότι έχουμε τον απαραίτητο χρόνο για συζητήσεις και συμφωνίες στο Συμβουλίο. Είμαστε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα των εκθέσεων και τη μετέπειτα ε, μελέτη τους από το Συμβούλιο. Ελπίζουμε ότι η εξέτασή τους την Άνοιξη θα προλιάνουν το έδαφος για πιθανές αποφάσεις στο Συμβούλιο του Ιουνίου. Αναγνωρίζουμε ότι είναι φιλόδοξο το θα είναι μεγάλη πρόκληση να το τηρήσουμε, ιδιαίτερα όταν λαμβάνω υπόψη μα του διάφορου παράγοντε που διέπουν τι αποφάσει μα. Μπορώ όμω να διαβεβαιώσω την Επιτροπή ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα εργαστεί επιμελέστατα για να κοιτάξει να διασφαλίσει πρόοδο σε σχέση με την πορεία προσχώρηση όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Πρέπει εδώ λοιπόν να επιβεβαιώσω ότι στηρίζει η Ιρλανδία και την προοπτική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Δεν ε, επίκυνται αποφάσεις από το Συμβούλιο για τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη επί προεδρίας μας. Ελπίζουμε όμως ότι οι επόμενοι μήνες θα δουν την ε, βοσνιακή κυβέρνηση και τους πολιτικούς ηγέτες να επιτελούν πραγματική και συνεχιζόμενη πρόοδο για να επιτύχουν τις ε, φιλοδοξίες της χώρας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η δέσμευσή μας αποδεικνύεται από την άτυπη συνάντηση υπουργών και υφυπουργών Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Δουβλίνο. Οι πέντε υποψήφιε χώρε ε, προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν και η συζήτηση αφιερώθηκε στη διεύρυνση. Επίση, ο Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η Υπουργό Λουσίντα Κρέιτον και ο Επίτροπο Φίλε συναντήθηκαν χωριστά με εκπροσώπου αυτέ τι τρει υποψήφιε χώρε για να συζητήσουν πώ θα ενθαρρύνουμε ε, τις χώρες αυτέ στην προσχώρηση. Επίση, ε, υπάρχουν τρει χώρε ήδη σε διαπραγματεύσει και συνεχίζεται η καθημερινή δουλειά για να προχωρήσει η διαδικασία επιστρέφω στην Κροατία, η οποία ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις και αναμένεται να προσχωρήσει την 1η Ιουλίου. Η Ιρλανδική Προεδρία θα ε, εποπτεύσει την ε, μελέτη για την ε, τελική μελέτη παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν θέματα υπομορφή σαφού καταλόγου εκκρεμών θεμάτων πρέπει να τα δούμε και όταν ολοκληρωθούν και αυτά θα είναι έτοιμοι για την προσχώρηση. Ισλανδία. Η Επιτροπή θα γνωρίζει τη συμφωνία μεταξύ του κυβερνητικού συνασπισμού ε, που θέλει να επιβραδύνει ε, τις διαπραγματεύσεις ε, για την προσχώρηση μέχρι τις εκλογές 27 Απριλίου. Όμως θα σημειώσατε επίσης και την πρόθεση συνεχιζόμενης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση επί των κεφαλαίων που είναι ανοιχτά ούτω ώστε να ε, ολοκληρωθούν και να κλείσουν. Η Ιρλανδία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την Ισλανδία προ αυτή την κατεύθυνση. Όλες οι υποψήφιε χώρε ε, έχουν βεβαίω το δικαίωμα να συνεχίσουν τι διαπραγματεύσει στο ρυθμό που εκείνες επιθυμούν και που θεωρούν κατάλληλο. Σεβόμεθα την απόφαση τη Ισλανδική κυβέρνηση, που καθ' όλη τη διαδικασία αυτή έδρασε με την μέγιστη δυνατή διαφάνεια σε όλε τι συναλλαγέ επί τη διαδικασία προσχώρηση. Η απόφαση αυτή κάπως μετριάζει τις αρχικές μας φιλοδοξίες. Όμως ελπίζουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ανοίξουμε δύο ακόμη κεφάλαια. Αυτά για τα οποία η Ισλανδία έχει ήδη υποβάλει διαπραγματευτικέ θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να κλείσουμε και τρία κεφάλαια. Η δέσμευσή μα θα συνεχιστεί με την Ισλανδία ο συνάδελφος υπουργό ε, για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις θα τα πάει στο Ρεκιάβη αύριο για περαιτέρω συναντήσεις. Τώρα, συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου για την Τουρκία να γνωρίζουν ότι είναι προς το συμφέρον των δύο μερών να, συνε... να... να ε, ε, αποκτήσουν πάλι δυναμική η διαπραγματεύση για την ένταξη. Η θετική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέτυχε να διατηρήσει την δέσμευση υπέρ της διαδικασίας. Οι τεχνικές ομάδες εργασίας που έγιναν σε κρίσιμους τομείς ε, συνεχίζονται ούτως ώστε να υπάρξει ευθυγράμμιση Τουρκίας ε, της νομοθεσίας με το κεκτημένο. Έχει προετοιμαστεί ένας ευρύτερος διάλογος και ένα πλαίσιο συνεργασίας με την Τουρκία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και οδικός χάρτης για καθεστώς χωρίς θεωρήσεις. Είναι σημαντικό τώρα η Τουρκία να υπογράψει παράλληλα τη Συμφωνία Επανεισδοχής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι προϋπόθεση για βήματα προς την απελευθέρωση θεωρήσεων ως σταδιακή και μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτές οι εξελίξεις κάθε έχουν μεγάλη αξία, αλλά δεν είναι υποκατάστατο για την καθ' αυτό πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Γνωρίζω ότι πέρασε αρκετός καιρός ε, από τότε που άνοιξε το τελευταίο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων το 2010 επί Ισπανική Προεδρίας. Ελπίζουμε να επιτελέσουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις επί δικής μας Προεδρίας και ελπίζουμε να ανοίξουμε τουλάχιστον ένα κεφάλαιο αν αυτό καταστεί δυνατό. Για να το επιτύχουμε θα στηριχθούμε στην προθυμία όλων των μερών και των κρατών μελών της Ένωσης και της Τουρκίας για να διευκολύνουμε την πρόοδο. Η Κυπριακή Προεδρία πέτυχε να ανοίξει το πρώτο κεφάλαιο διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο. Καθώς συνεχίζεται η διαδικασία ε, εξέτασης, ε, screening, ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουμε και θα ανοίξουμε άλλο ένα κεφάλαιο, ίσως και δύο. Το διαπραγματευτικό πλαίσιο και το Μαυροβούνιο δείχνει τη νέα προσέγγιση η οποία ε, βλέπει πρόοδο ε, σε ε, θέματα που αφορούν δικαιοσύνη και συνδέεται με άλλα θέματα. Ολοκληρώθηκε η εξέταση αυτών των κεφαλαίων, θεμελιώδη δικαιώματα, δικαστικό σώμα, δικαιοσύνη, ελευθερία, ασφάλεια. Ε, το προσκλήθηκε για το Μαυροβούνιο να συμμετέχει στο προγράμματα δράση, τα οποία είναι η, τα πρώτα ε, ορόσημα συγκριτική αξιολόγηση αυτά τα κεφάλαια. Οπωσδήποτε θα δώσουμε χρόνο γιατί χρειάζεται, αλλά ενθαρρύνομαι προ αυτή την κατεύθυνση την πρόοδο. Τέλος, ε, για τη διεύρυνση. Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας λέει ότι το 2013 η Ιρλανδική Προεδρία θα συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα σε αξιόπιστη πολιτική διεύρυνση με βάση την αρχή της ε, αιρεσιμότητα, ε, Αξιόπιστος, αξιοπιστία και αιρεσιμότητα, πολύ σημαντικό. Η αιρεσιμότητα είναι σημαντική στην διαδικασία διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση, είναι σημαντικό να παραμείνει αξιόπιστη διαδικασία. Έτσι οι προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι αυστηρές, ούτω ώστε να είναι βέβαιο ότι οι προσχωρούσες θα είναι απόλυτα προετοιμασμένες και θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες της, ε, του μέλους. Παράλληλα, θα πρέπει να παραμείνουν αξιόπιστε και επιτεύξιμες οι προϋποθέσεις και δεν θα πρέπει να γίνουν μη ρεαλιστικέ, ούτω ώστε να παρεμποδιστούν οι χώρες από το να ακολουθήσουν την οδό τη Εντάξει, η Ιρλανδική Προεδρία ε, δίνει μεγάλη έμφαση σε μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα στοχεύσουμε για να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις στις επόμενους, τους επόμενους μήνες. Η προσχώρηση είναι περίπλοκη διαδικασία, δύσκολη, απαιτητική. Αναμφίβολα οι νέες υποψήφιες χώρες θα κρυθούν πιο αυστηρά από ότι οι προκάτοχή τους. Ε, μεταξύ άλλων λόγω της διεύρυνσης ε, και της εμπάθυνσης του κεκτημένου. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική στη διαδικασία και ελπίζω να τα καταφέρουμε στην Προεδρία μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται συχνά ως η φωνή του λαού. Όταν μιλάμε για την πολιτική διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η υποστήριξή σα είναι ζωτική, γιατί διασφαλίζει ότι τα, οι ανησυχίε των λαών τη Ευρώπη και των πολιτών και ε, των χωρών μελών και των υποψηφίων θα εισακούονται. Και οι αλλαγέ, οι πρόοδοι, τα ωφέλη από την πολιτική θα ε, κοινωνούνται στου λαού με την υποστήριξή σας είμαι σίγουρος ότι η διεύρυνση θα παραμείνει μια αξιόπιστη πολιτική ισχυρή που θα συνεχίσει να ωφελεί τους πολίτες των χωρών της διεύρυνσης και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζει η συζήτηση, πολλές είναι οι ερωτήσεις και λίγος ο χρόνος. Γι' αυτό θα πρέπει να κάνετε σύντομες παρεμβάσεις. Δύο λεπτά το πολύ. Η κυρία Γκόμες θα δώσει το πρώτο παράδειγμα. Καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ. Δεν πρέπει να περιοριστούμε στη διεύρυνση, έτσι δεν είναι. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Μιλάτε για σταθερότητα, ανάπτυξη και απασχόληση. Υποφέρουμε στην Ευρώπη σχετικά. Έχουμε τεράστια φοροδιαφυγή, για παράδειγμα. Εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι για να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή συνολικά και για τις υπονάπτυξη χώρες που επίσης υποφέρουν από αυτό το φαινόμενο μπορείτε να κάνετε κάτι. Έπειτα έχουμε την πρόκληση να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας σχετικά με την, το Μαλί και την ασφάλεια εκεί. χώρες όπως είναι η δικιά σας και η δικιά μου. Πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να συνεισφέρουν ε, περισσότερο αν υπάρξει ενίσχυση στα οικονομικά. Η κυρία Νέης. Πρόεδρε. Αυτό που είπε η κυρία Γκόμες με κάνει να πάω λίγο πίσω στην εποχή του Μακιαβέλη όπου είχαμε σχόλια για τα θετικό ή αρνητικό του να χρησιμοποιεί κανείς τους δικούς του στρατιώτες ή τους ξένους και λέγανε ότι άμα χρησιμοποιείς τους δικούς στρατιώτες είσαι πιο αποτελεσματικός. Τέλος πάντων, αυτό είναι παράπλευρο. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Χτες το απόγευμα και σήμερα ε, συζητούσαμε τις διάφορες εκθέσεις πρόοδου σχετικά με τις υποψήφιες χώρες. Ορισμένες όπως η Κροατία είναι περίπου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες βρίσκονται στο προφάλαμο της όλης διαδικασίας. Και μπορώ να πω ότι η δικιά μου η αντιπροσωπεία συμφωνεί με την προσέγγιση που μας παρουσιάσατε σήμερα και τη φιλοδοξία της Ιρλανδικής Προεδρίας. Μια ερώτηση έχω. Μάθαμε με πόνο ότι δεν είναι καλή ιδέα να δεχόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία χώρα η οποία όμως έχει πρόβλημα σε εκκρεμότητα με μια γείτονα χώρα ή με κάποια άλλη, εν ότι δεν βοηθάει. Όταν υπάρχει λοιπόν μια υποψήφια χώρα που έχει ένα άλλο το πρόβλημα με μια χώρα μέλος, εσείς αναφερθήκατε σε διάφορες χώρες που θα μπορούσαν να θελήσουν να τους απονεμηθεί το καθεστώς της υποψήφιας χώρας, αλλά ότι είναι εμπλεγμένες σε διάφορες παγωμένες διαμάχες με γείτονές τους χώρες. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, γιατί εμείς ως Κοινοβούλιο πάντα προσπαθούσαμε να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Δηλαδή, να μην αφήσουμε οι χώρες που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν όμοιροι των άλλων χωρών με τις οποίες έχουν διαμάχη. Αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να βάλουμε και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια χώρα με ένα άλλο το πρόβλημα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει παρεντέρω προβλήματα. Η δικιά σας η άποψη ποια είναι γι' αυτό. Ο κύριος Σκύλαν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για το δυναμισμό σας, την πεποίθησή σας και την ρεαλιστική σας παρουσίαση. πρόκειται για μια συμμετρική ή ασύμετρη προσέγγιση, γιατί εσείς δεν αναφερθήκατε καθόλου στην ανατολική διάσταση της Ευρώπης. Η ασυμμετρη προσεγγιση γιατι εσεις δεν αναφερθηκατε καθολου στην ανατολικη διασταση της ευρωπης η πολιτικη ε, για την ε, ετορική σχέση ανατολικά ε, είναι κάτι που δεν αναφέρατε. δικιά σας η προσέγγιση ποια είναι. Είσαστε φιλόδοξος. Ουκρανία, Μολδαβία, Λευκορωσία μια προσχώρησή του η στενή συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς σας βρίσκει. Και πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάποια σημαντική αλλαγή για το θέμα της Μακεδονίας. Έχει καθυστερήσει πολύ, για χρόνια. Και νομίζω ότι εσείς έχετε μπροστά σας μια εξαίρετη ευκαιρία να λύσετε αυτό το ζήτημα. Ε, κυρία σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Υπουργό Γκίλμορ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ επίσης για τα όσα είπατε, για αυτά τα οποία θέλετε να πετύχετε κατά τη διάρκεια της εξάμενης Ιρλανδικής Προεδρίας για τη διεύρυνση. Μας πεθυμίσατε το 2004 όταν μπήκαν 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήσασταν εσείς στην Προεδρία. Θυμάμαι την ημέρα αυτή, ήταν μια μέρα μεγάλης ευτυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μολονότι υπήρχαν τότε προβλήματα με κάποιες χώρες και με κάποιες που ακολούθησαν μετά. Μετά από αυτά που είπε η προτείναμε νομίζω σε ένα από το ψήφισμά μας που συζητήσαμε χθε ή σήμερα, δεν θυμάμαι πολύ καλά πλέον, είπαμε πάντως ότι θα πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός διαμεσολάβησης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι χώρες οι οποίες εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να εμποδίσουν άλλες χώρες να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας διμερών τους διενέξεων και προβλημάτων. Σας έχει απασχολήσει αυτό, θα το συζητήσετε αυτό με τους συναδέλφους σας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κατανομάσουμε αυτή τη στιγμή χώρε. Το πρόβλημα υφίσταται, συσσωρεύονται προβλήματα στο παρελθόν και νομίζω ότι τέτοια προβλήματα θα έχουμε και στο μέλλον. Πώ θα προσεγγίσετε ουσιαστικά το ζήτημα αυτό να προβλεφθεί, προβλεφθεί ένα τέτοιο μηχανισμό. Επίση, κύριε Υπουργέ, Είπατε ότι θέλετε να σημειωθεί πρόοδος για την Σερβία και το Κωσυφοπόδιο, στη μεταξύ, Κωσυφοπέδη με συγχωρείτε, στη μεταξύ τους, στο μεταξύ τους διάλογο. Εγώ είμαι εισηγήτρια για το Κωσυφοπέδιο, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όντως το Συμβούλιο να πει το τελικό ναι προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σύνδεσης και σταθερότητας πριν το καλοκαίρι. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι ενδιασμοί από ορισμένα κράτη-μέλη όσον αφορά το καθεστώ του κοσφοπεδίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει πει όμω ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία νομική πτυχή η οποία θα εμπόδιζε μία τέτοια διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας. Εσείς πώς βλέπετε την κατάσταση, αν το κοσφοπέδιο τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις, ως Ιρλανδική Προεδρία θα πιέσετε προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης και Σταθερότητας με το κοσφοπέδιο και σε σχέση με αυτά που είπε η Άννα Γκόμες κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με την διεύρυνση όσο πολύ, αλλά με τη γενικότερη εξοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λήφθη μια απόφαση για 11 χώρες όσον αφορά το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Θα ζητούσα και από τη δική σας την κυβέρνηση να μην συνεχίσει να προωθεί αυτή τη χαμηλή εταιρική φορολογία που υπάρχει στην Ιρλανδία. Νομίζω ότι δεν βάζεται ένα καλό παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Δεν θέτετε εσείς ένα θετικό παράδειγμα για τις χώρες της διεύρυνσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Λέει ο κύριο Τάνοκ, πολύ θετικό το παράδειγμα το οποίο έχει δώσει η Ιρλανδία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τις προτεραιότητές σας. Μιλήσαμε για τα Δυτικά Βαλκάνια σήμερα. Βλέπω ότι είστε και υπουργό Εμπορίου. Ξέρετε ότι στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να βγει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να μπορεί η χώρα μου ελεύθερα να διαπραγματεύεται εμπορικά με τον υπόλοιπο κόσμο. Μα η παρουσία τη Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε καμία περίπτωση δεν την εμπόδισε να διαπραγματεύεται ελεύθερα με τον υπόλοιπο κόσμο. Και νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθηθεί περισσότερο ακόμα και από κάποιους Αμερικανούς ηγέτες για το πώς τελικά ανοίγεται προς την υπόλοιπο κόσμο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν οι 27 Υπουργοί Εμπορίου να καταφέρουν τελικά να πετύχουν μια καλύτερη συμφωνία εμπορική από ότι αν κάθε χώρα διαπραγματευόταν ξεχωριστά. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προωθήσουμε πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να δοθεί και ως μάθημα στον Ομένο Βασίλειο που θέλει να δράσει μονομερός. Σας ε, ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε κύριε Γκίλμορ. Είμαι εισηγητής ε, για την Μακεδονία. Ξέρω ότι ε, υπάρχουν οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε μία σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών. Πάντως, ο Επίτροπος Φούλε έκανε κάποιες προτάσεις, αλλά από ό,τι φαίνεται όμως τα κράτη-μέλη στα πλαίσια του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή έχουν διστάμενες απόψεις. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει όμως να επαναληφθεί αυτό στο μέλλον. Η απογοήτευση θα είναι τεράστια και θα περάσουν πάλι πάρα πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρει η Μακεδονία να ξεκινήσει πάλι την όλη διαδικασία της προσέγγισής της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πολλοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούν ότι ε, πρέπει και το Συμβούλιο να συμβάλλει πολύ σημαντικά από διπλωματικής πλευράς να ασκήσει πίεση στα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλήξει μέχρι τον Ιούνιο το Συμβούλιο σε μια θετική συμφωνία. Υπάρχει το ζήτημα της ονομασίας, το οποίο δεν πρόκειται δυστυχώς να λυθεί μέχρι τον Ιούνιο. Ασκούμε πίεση γι' αυτό. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι αν δεν συμβεί τίποτα, τα πράγματα θα είναι πολύ επιζήμια. Προσπαθήσαμε επίσης να προωθήσουμε αλλαγές ε, όσον αφορά τη στάση των ε, αρχών της Μακεδονίας για την αλβανική μειονότητα. Ξέρετε ότι ε, έχουν συναυθεί πολλές συμφωνίες με το Κωσυφοπαίδιο. Ξέρετε πόσο αυτό συνέβαλε στο να προωθηθούν οι σχέσεις Κωσυφοπαιδίου και Σερβίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε όλες αυτές τις αλλαγές που γίνονται στα Δυτικά Βαλκάνια να μην απομονωθεί η Μακεδονία. Δεν μπορούμε να εμείνουμε αυτή τη στιγμή στην υφιστάμενη κατάσταση, στο status quo. Ξέρω ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία έχουν θεμητούς λόγους να αντιδρούν και έχουν θεμητές ενδια... Ε, ενδιασμούς, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεχομένω να μην καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Γι' αυτό το λόγο σας ζητώ να χρησιμοποιήσετε όλες τις διπλωματικές σας δεξιότητες προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία στο Συμβούλιο. Σας υποστηρίζουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, καλωσορίζω και εγώ τον ε, ε, Υπουργό Εξωτερικών και Εμπορίου της Ιρλανδίας. Θα ήθελα με την ευκαιρία της παρουσίας του να αναφερθώ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ε, στρατιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω αν θα έχουμε σύντομα τη δυνατότητα να μιλήσουμε τα ζητήματα αυτά. Δύο ερωτήσεις έχω να σας κάνω κύριε Υπουργέ. Η πρώτη ερώτηση ε, αφορά την υπεριαλιστική επέμβαση της Γαλλίας στο Μαλί και η ερώτησή μου η συγκεκριμένη είναι τι μέτρα θα πάρετε εσείς ως Προεδρία να σταματήσει αυτός ο απαράδεκτος πόλεμος ο οποίο γίνεται για πρώτε ύλε και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που επικαλείται η γαλλική κυβέρνηση. Δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με το πολύ βαρύ πρόγραμμα τη ε, Ιρλανδική Προεδρία όσον αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα και θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Η Ιρλανδία είναι μια ουδέτερη χώρα. Αυτό θέλει ο λαό τη, αυτά προβλέπουν οι μέχρι τώρα καταστάσει. Δεν βλέπετε να υπάρχει μια ε, διαφωνία, μια αντιπαράθεση, μια αντίθεση μια αντίθεση, αυτός, αυτός είναι ο σωστός όρος, μεταξύ της ευθύνη σας να διαχειριστείτε πολέμους όπως είναι αυτός του Μαλή, ενδεχομένως της Συρίας, αλλά κυρίως το πρόγραμμα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, δεν υπάρχει μια αντίθεση με το στάτους της ουδετερότητας της χώρας σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε ως πρώην υπουργό στην Ιρλανδία. Φόρεσα την ειδική μου ε, γραβάτα ε, του ε, οπαδού του ποδοσφαίρου. Ο Τίσοκ συνόψισε την ε, συζήτηση ακολουθώντας πιστά τις μεγάλες παραδόσεις του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να ε, υπενθυμίσω κάτι που είπε και ελπίζω να το μεταφέρετε. Το τελευταίο που θέλετε είναι να είστε υπουργό μιας μείωσης μαζί με τον κύριο Τάνοκ πιστεύω και ελπίζω και εγώ ότι θα κάνετε ότι είναι δυνατόν ως μεγάλος φίλος του Ηνωμένου Βασιλείου για να διασφαλίσετε ότι ο Βρετανικός λαός θα καταλάβει ότι καλύτερα είναι μέσα παρά έξω. Και τέλος, ε, να σας ρωτήσω κάτι άλλο, δεν αφορά την διεύρυνση τόσο πολύ. Ε, οι Ισραηλινές εκλογές είναι πολύ σημαντικές. Ε, ξέρω ότι έχετε πάει στη Γάζα. Ε, γιατί ε, ε, σας παρακολούθησα το πρόγραμμά σας, ξέρω τα προβλήματα που είχατε. Μπορείτε να δώσετε σημασία στο θέμα το Παλαιστινιακό μετά τις εκλογές του Ισραήλ, γιατί φαίνεται ότι παίρνει πάλι πολύ επικίνδυνες και καταστροφικές διαστάσεις. Και να σας ευχηθώ ότι καλύτερο για το εξάμεινο της Προεδρίας σας. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε, είμαι Σλοβάκος ε, από μία από τις δέκα χώρες που προσχώρησαν επί προεδρία σας το 2004 και θυμόμαστε την εξαιρετική προεδρία και την καταπληκτική υποδοχή στο Κόρκο που μας υποδεχθήκατε τότε. Εκτιμώ το γεγονός ότι μετά από μακρές συζητήσεις για κάθε χώρα στα Βαλκάνια σχετικά με την φιλοδοξία ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, αποδίδεται μεγάλη σημασία, προσέχετε πολύ και μας αναφέρετε συγκεκριμένα τα σχέδιά σας για κάθε χώρα της περιοχής. Ξέρω ότι είστε ρεαλιστές προσγειωμένοι άνθρωποι που προτιμάτε τα μικρά αποτελέσματα παρά τα ε, μεγάλα σχέδια που είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Μια και μιλούσαμε για κάθε μια από τις χώρες στην περιοχή, ενθαρρύνομαι να ρωτήσω, γιατί το όνομα Αλβανία νομίζω το αναφέρατε, αλλά ξέχασα αν προσθέσατε κάτι. Ε, και εκείνοι ε, ε, και οι υποψήφιες χώρες περιμένουν με ενδιαφέρον. Το Ιούνιο εκεί θα γίνει η επιπροεδρία σας ακόμα, θα γίνουν εκλογές στη χώρα. Τι ελπίδα ρεαλιστική όμως μπορείτε να προσφέρετε σε αυτή τη χώρα. Thank you. Minister. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, δεν χρειάζεται να σας ε, επαναλάβω ότι οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες στηρίζουν τους συνολικούς στόχους της Ιρλανδικής Προεδρίας και συγκεκριμένα την πολιτική για την ε, διεύρυνση. Δεν θα μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες γιατί εσείς τις αναφέρατε. Θα ήθελα μια προσέγγιση πολιτική και οικονομική περισσότερο. Γιατί αν δούμε χώρες όπως τη Σερβία ή τη Μακεδονία ή την Αλβανία, αυτές οι χώρες είναι χώρες φτωχές. Δεν έχουν οικονομική ανάπτυξη, έχουν υψηλότατη ανεργία και οι, χώρες, οι, εταιρείες μας αντί να επενδύουν στις χώρες αυτές σε φαντουργία, ένδυση κλπ. Προτιμούν να επενδύσουν στην Κίνα όπου η, ε, εντωμεταξύ η μισθή είναι υψηλότερη από τη Σερβία και την Μακεδονία και μετά εξάγουν τα εμπορεύματά τους ε, στην Ευρώπη και στις χώρες της Ένωσης. Θα είχε λοιπόν νόημα και ε, εμπιστεύομαι την, ότι η Ιρλανδική Προεδρία τουλάχιστον θα ανοίξει τη συζήτηση από αυτού του θέματος ε, για να υπάρξει βιομηχανική πολιτική, μέτρα για τη βιομηχανία και σε εμά και στις γειτονικέ χώρες που θα έχουν πολιτικό και οικονομικό νόημα, ούτω ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη, να ε, ε, δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας σε χώρες όπως η Αλβανία, η Σερβία, η Μακεδονία. Μην εστιάζουμε μόνο στα τεχνικά θέματα, δηλαδή στα κεφάλαια και στα ορόσημα συγκριτικής αξιολόγησης, αλλά να ε, έχουμε την πολιτική και την οικονομία υπόψη μας, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε και τις χώρες της διεύρυνσης και τα κράτη-μέλη επίσης. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Τουρκία. Σωστά είπατε ότι η Προεδρία θέλει να προχωρήσει την διαδικασία τα το τραύμα των τελευταίων μηνών υπό την προηγούμενη Προεδρία, την Κυπριακή. Σωστά. Όμως δεν περιμένουμε και θαύματα, ουσιαστική πρόοδο δεν φαίνεται να υπάρξουν αλλαγές στην τρέχουσα διαδικασία παρά τα όσα είπε ο κύριος Ολόντ. Όμως υπάρχει πρόοδος και είναι ζωτική σημασία να το αναγνωρίσουμε αυτό πρόοδος στο κουρδικό. Η τουρκική δημοκρατία και το ΠΚΚ απέτυχαν και οι δύο να λύσουν το κουρδικό ζήτημα. Όμως η αλλαγή είναι, η πρόοδος είναι ότι το έχουν αντιληφθεί πια αυτό και οι δύο πλευρές. Και οι συνομιλίες με τον κύριο Τσαλάν και την κυβέρνηση είναι ένα μήνυμα για μια νέα αρχή. Και μια νέα αρχή μπορεί να στηριχθεί και να εθαρρυνθεί από μας και θα έπρεπε. Ελπίζω, αν έχετε την ευκαιρία να βγείτε λίγο από τα αναγκαία, τα τυπικά, τους περιορισμούς που έχει βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορείτε λοιπόν καλό θα ήταν να στείλετε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα στην Άγκυρα που να λέει ότι μπορεί να υπάρξει φρέσκος αέρας που να μπαίνει στη διαδικασία όσον αφορά το κουρδικό ζήτημα και ότι αυτό το στηρίζουμε εμείς πολιτικά και ηθικά. Ο Υπουργό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Το θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η διεύρυνση, είχα καταλάβει, αλλά οι ευρωβουλευτές εδώ το ερμηνεύουν ε, πιο έτσι ανοιχτά. Και διεύρυναν και την ημερήσια διάταξη επιτυχώς. Θα απαντήσω με τη σειρά στα διάφορα ζητήματα. Κυρία Γκόμες το θέμα της διαφθοράς. Φυσικά και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αντιμετωπίσει το θέμα της φοροδιαφυγής. Με συμμόρφωση στις διάφορες συμφωνίες. Ρωτήσατε πιο συγκεκριμένα για το Μαλί. Οι προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να πιέσουμε τους πολιτικούς ηγέτες στο Μαλί να προχωρήσουν για την αποκατάσταση του ε, νόμου δικαίου. Επικεντρωνόμαστε σε θέματα διαιτησίας και ετοιμάζουμε μια νέα ευρωπαϊκή αποστολή κατάρτιση εκεί του στρατού και της αστυνομίας και βέβαια φροντίζουμε και η ανθρωπιστική βοήθεια. Και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει και πάλι συνεργασία σε επίπεδο ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση. Σίγουρα τα κράτη-μέλη είναι αυτά που χρηματοδοτούν. Δουλεύουμε και πάνω στην κοινή χρηματοδότηση και θέλουμε να υπάρξει μια ισορροπία εκεί. Κυρία Νέιτς. Το θέμα των διμερών ζητημάτων. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται για την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνονται με συνένεση. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Όταν συζητάμε τόσο βασικά ζητήματα όπως είναι το κατά πόσο μια χώρα θα γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Είναι σημαντικό να κοιτάμε όλες τις παραμέτρους και την αξιοπιστία της διαδικασίας βέβαια προσχώρησης και φυσικά και πρέπει να εξετάσουμε θέματα όπως είναι αυτά, οι διμερείς διαφορές τις οποίες αναφερθήκατε. Και πρέπει να το πούμε ότι η διαδικασία της διεύρυνσης η ίδια είναι, το έχουμε δει τόσες φορές στο παρελθόν, είναι μία διευκόλυνση, μία ενθάρρυνση για τη λύση τέτοιων διμερών διαφορών. Κύριε Κίλαμ, για το θέμα της εταιρικής σχέσης με τις ε, χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν ανέφερα τίποτα, αλλά θα σας πω για να χαρείτε ότι χτες, χτες Δευτέρα, ναι, έχω μπερδέψει και τις μέρες, χτες λοιπόν είχα την ευκαιρία να συζητήσω με τον Λιθουανό συνάδελφο που ήταν στο Δουβλίνο για ένα τυπο συμβούλιο και το θέμα αυτό συζητήθηκε. Ξέρουμε ότι έχει προχωρήσει από τον Νοέμβριο. Οι διάφορες προεδρείς συνεχίζουν την ίδια πορεία. Συζητάμε λοιπόν την προοπτική συνεργασίας με την Ουκρανία, τη Μολδαβία, Λευκορουσία κτλ. Και παρατηρούμε και τις προετοιμασίες που κάνει η Λιθουανία για να ετοιμάσει την επόμενη συνάντηση. Όσον αφορά την τέος Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας τώρα. Και ο κύριος Χαουβιτ αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, χαιρόμαστε με τα συμπεράσματα που καλωσορίζουν την έκθεση πρόδου για διάφορα σημεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο φυσικά με το διάλογο υψηλού επίπεδου για την προσχώρηση. Οι αρχές της ΦΥΡΟΜ έχουν προχωρήσει αποφασιστικά στις μεταρρυθμίσεις το Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άνοιξη του 2013 να ενημερώσει για την πρόοδο των παρετέρω μεταρρυθμίσεων. Περιμένουμε λοιπόν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από εκεί και πέρα εμείς θα προωθήσουμε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την ΦΥΡΟΜ εφόσον το Συμβούλιο το αποφασίσει. Γίνονται αποφάσεις, όπως είπαμε και πριν, με ομοφωνία όσον αφορά την προσχώρηση νέων χωρών η Ιρλανδία ως προεδρεύουσα χώρα και όπως είπατε θα ε, φροντίσει να προωθήσει το θέμα και να συζητηθεί μετά βέβαια την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε συμφωνία για αυτό το θέμα. Φυσικά θα παρατηρούμε προσεκτικά τι γίνεται, ιδιαίτερα μάλιστα τις συζητήσεις στη Νέα Υόρκη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα του ονόματος. Κυρία Λούνατσεκ. για το θέμα των ε, μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να μπλοκάρουν, να εμποδίσουν αποφάσεις διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσχώρησης δηλαδή ενός νέου μέλους. Το πρώτο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πρέπει να σεβόμαστε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τις προωθούμε. Και αυτό πρέπει να φαίνεται ότι το φροντίζουν όλες οι υποψήφιες χώρες. Πιστεύω επίσης, ξέρετε η διαδικασία διεύρυνσης, όπως σας είπα πριν, πρέπει να είναι αξιόπιστη. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη ατζέντα με σχετικά με τη διεύρυνση και πρέπει να την προχωρήσουμε. Αλλά όπως λέτε δεν πρέπει ένα μεμονωμένο μέλος να εμποδίζει τη συνέχεια της διαδικασίας αυτής. Ε, συμμερίζομαι και εγώ, μια που είσαστε εισηγήτρια για το κοσυφοπαίδιο, συμμερίζομαι και εγώ τις ε, απόψεις σας και ελπίζω να ανακουφιστούμε λίγο από τη θετική γλώσσα που ακούμε από την ηγεσία του Βελιγραδίου. Η Ιρλανδία δεν είναι μια χώρα χαμηλών φόρων. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι αποτελεσματικά ε, επίπεδα φορολόγησης στη μέση θα έλεγα ότι είμαστε σε σχέση με τις υπόλοιπε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εντάξει, αυτό θα το συζητήσουμε παρετέρω κάποια άλλη στιγμή. Μη σπαταλάω το χρόνο σας. Για τον κύριο Τάνοκ τώρα. Και τον Σερόμπερτ. Ρόμπερτ. Μου ζητήσατε τη γνώμη μου σχετικά με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για τη σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιρλανδία έχει φάει τόσο χρόνο να ακούει από το Ηνωμένο Βασίλειο τι πρέπει να κάνει, που όπως καταλαβαίνετε ε, δυσκολεύομαι να το αντιστρέψω αυτό και να αρχίσω εγώ να λέω στο Ηνωμένο Βασίλειο τι θα πρέπει να κάνει. Αλλά κοιτάξτε τώρα για τις εμπορικές συμφωνίες. Εκεί Σίγουρα θέλουμε να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας, οπότε τι έχω να σας πω γι' αυτό. Ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και μπορούμε να έχουμε εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία και με τους άλλους στρατηγικής σημασία εταίρους μας που προσθέτουν 2% στο ευρωπαϊκό ΕΠ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, είμαστε συλλογικά πολύ πιο δυνατοί, πολύ καλύτεροι, πολύ πιο έτοιμοι να κερδίσουμε τις εμπορικές αυτές συμφωνίες όλοι μαζί, μια που πρόκειται για 500 εκατομμύρια ανθρώπους, τεράστια αγοραστική δύναμη, φυσικά και είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση, άπαξ και διαπραγματευόμαστε εμπορικέ συμφωνίε όλοι μαζί, συλλογικά ω Ευρωπαϊκή Ένωση, από ότι μεμονωμένο ο καθένα μα. Είτε είμαστε μια μικρή χώρα, είτε είμαστε μια μεγάλη χώρα. Η Ιρλανδία, το είπα στην αρχή στην παρουσίασή μου, ότι 40 χρόνια τώρα είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά είναι και 40η επέτειος προσχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαζί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε και έχουμε αναπτυχθεί μαζί για διάφορα θέματα, εμπόριο, ενιαγορά. Ένα σωρό θέματα που συζητήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια εδώ μαζί στον ίδιο δρόμο βρισκόμασταν το Ηνωμένο Βασίλειο και εμείς. Είμαστε και γείτονε και πολύ καλοί φίλοι σήμερα. Έχουμε από κοινού ευθύνη για την ειρηνευτική διαδικασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και το έχω πει δημόσια και το επαναλαμβάνω ότι η Ιρλανδία θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο να είναι ένα πλήρες δεσμευμένο υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέλος μέσα σε αυτήν. Νομίζω ότι είναι καλύτερο αυτό για όλους όχι μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στον κύριο Αγκουράκη τώρα. Σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε σε σχέση με την Ιρλανδία που είναι ουδέτερη χώρα. Ναι, είμαστε ουδέτερη χώρα, δεν συμμετέχουμε σε στρατιωτικούς συνασπισμούς. Είναι μέρος του συνταγματός μας αυτή η δέσμευση. Όμως το ότι είμαστε ουδέτερη χώρα δεν σημαίνει ότι παίρνουμε τις αποστάσεις μας ή μπαίνουμε στην πάντα και δεν ασχολούμαστε με τα σημαντικά θέματα. Κανένας δεν μπορεί να κάνει στην πάντα. Για αυτά που συμβαίνουν στη Συρία, τη σφαγή των ανθρώπων, 60.000 άνθρωποι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους. Ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, με το οποίο ασχολείται το Συμβούλιο και η ε, εκπρόσωποι. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε, επειδή είμαστε ουδέτεροι. Τρομοκρατία έπειτα. Ε, μαλλί ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε από αυτό μπορούμε να πάρουμε αποστάσεις και να παραμείνουμε αδιάφοροι. Το ότι είμαστε ουδέτερη χώρα δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για πράγματα τα οποία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Για το θέμα της Αλβανίας. Ο κύριος Κούκαν αναφέρθηκε σε αυτό. Α, όχι, σε αυτό θα έρθω σε λίγο. Κύριε Νταφ, πρώτα, Τουρκία. Νομίζω ότι είναι σωστό να πούμε πως το θέμα της τουρκικής προσχώρησης, ένταξης, είναι κάτι που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δυόμιση χρόνια τώρα έχουμε κολλήσει κάπως, όχι μόνο τους τελευταίους έξι μήνες υπό Κυπριακή Προεδρία, εγώ ελπίζω να ανοίξει και κάποιο ακόμα κεφάλαιο κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας χάρη στο δυναμισμό που θα αποκτήσει και πάλι η διαδικασία. Σίγουρα παραμένουν πολλά ζητήματα που πρέπει να προχωρήσουν. Ο Τούρκος υπουργό ήταν πριν τα Χριστούγεννα στην Ιρλανδία και είχαμε μια καλή συζήτηση για κάποια από τα ζητήματα που πρέπει να προχωρήσει η ίδια η Τουρκία. Υπάρχουν και πολλά πολιτικά ζητήματα βεβαίως που πρέπει να λύσει η Τουρκία, όπως αυτά που αναφέρατε. Και ναι, πρέπει να στέλνονται πολιτικά μηνύματα. Τώρα, κύριε Κούκαν για την Αλβανία. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι πρέπει να συγχαρούμε την Αλβανία για την πρόοδο που πέτυχε με τις μεταρρυθμίσεις που θέτησε τον τελευταίο καιρό. Όμως το συμπέρασμα είναι ότι ακόμα μένουν μέτρα να ληφθούν πριν αποκτήσει το ε, καθεστώς της υποψήφιας χώρας, θέματα μεταρρύθμισης της διοίκησης και άλλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κληθεί να αναφέρει στο Συμβούλιο όταν έχει επιταχθεί επαρκή πρόοδο και το Συμβούλιο βέβαια θα αποφασίσει αν θα πάρει η Αλβανία το καθεστώς της υποψήφια χώρας ή όχι. Πρέπει πρώτα να έχουμε θετική έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει και ότι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο υπό τις Προεδρίες μα. Τέλο, κύριε Ρούτσεκ. Αυτό που είπατε Κοιτάξτε, μιλάμε για τη διεύρυνση και μπορούμε να μιλήσουμε πολύ τεχνικά, να αναφερθούμε στα κεφάλαια, στις εκθέσεις, τεχνικά ζητήματα που αναλαμβάνουν βέβαια οι ειδικοί μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αξιωματούχοι του Συμβουλίου και οι δικοί μου συνεργάτες στο Δουβλίνο και στις Βρυξέλλες. Αλλά ως πολιτικοί, γιατί είμαστε πολιτικοί όλοι εμείς εδώ πρέπει να θυμόμαστε ότι ο λόγος που τα κάνουμε όλα αυτά είναι το συμφέρον του κόσμου. Είναι οι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη σημερινή και οι άνθρωποι οι πολίτες των υποψήφιων χωρών. Όσον αφορά τους λόγους της Ευρώπης, είναι η οικονομία πολύ βασικό. Είναι η απασχόληση του τους ενδιαφέρει. Είναι το επίπεδο ζωής τους. Σταθερότητα, απασχόληση και ανάπτυξη. Σας είπα ότι αυτό είναι το μότο μας. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ασχοληθήκαμε με τις τράπεζες, τα δημοσιονομικά και όλα τα σχετικά. Αλλά εκπροσωπούμε τους λαούς μας και οι κυβερνήσεις μας, αλλά πολύ περισσότερο εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο, πρέπει να ξέρουμε ότι οι άνθρωποι περιμένουν από εμά να υιοθετούμε αποφάσεις οι οποίες να έχουν νόημα για αυτούς. Ότι θα έχουν καλύτερη δουλειά, ότι τα παιδιά τους θα έχουν καλύτερο μέλλον, θα βελτιώσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες, την ε, εκπαίδευση κλπ. κλπ. Ότι το μέλλον τους θα είναι καλύτερο και ότι δεν θα δέχονται απειλές περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει το Κοινοβούλιο. Ότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για τον κόσμο. Είτε το κάνουν οι κυβερνήσει των χωρών μελών, είτε το κάνουν οι αξιωματούχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να γίνεται για το συμφέρον του κόσμου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για τη συζήτηση αυτή, για την ομιλία σας, για τις δεσμεύσεις σας. Έχω τη θετική αίσθηση ότι θα έχουμε πραγματικά μια πολύ επικοδομητική συνεργασία τους επόμενους έξι μήνες. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας, γιατί δική σας επιτυχία θα είναι και δική μας επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.